Right. Can I have your attention, please? Uh, my pleasure to welcome you to the meeting this afternoon. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας συνεδρίαση. Προσπάθησα να ξεκινώ όσο δυνατόν πιο νωρίς. Ξέρω ότι έχουμε κάπως καθυστερήσει, αλλά επισημαίνω ότι στις 5 θα πρέπει να σταματήσουμε σήμερα, καθώς έχουμε μια άλλη συνεδρία σε μεικτή αυτή τη φορά. Ε, θα είμαστε όσο δυνατόν πιο αυστηροί λοιπόν στο ε, πρόγραμμά μας για να τηρήσουμε τον χρόνο. Και ξεκινώντας, ζητώ συγγνώμη ε, εκ μέρους του κ. Βαρτρή, ο οποίος μόνο στις 4.30 θα μπορέσει να φτάσει, καθώς είχε υποχρεώσει ανελειμμένες στην Γαλλία. Θα έρθει το χειρότερο δυνατό λοιπόν. Και Περνώ στην έγκριση της ημερησίας διατάξεως, επισημένοντας ότι το σημείο 17 μας ζητήθηκε να έρθει πιο νωρίς. Η κυρία Χολμάιερ θα έρθει σε λίγο και άρα θα το δούμε μετά το 9. Αύριο το πρωί. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις μετά το 9, αύριο το πρωί το σημείο 17. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Και επαναλαμβάνω ότι έχουμε πίεση χρόνου και θα τηρήσουμε στο δυνατόν πιο αυστηρά το πρόγραμμα μας. Αύριο το πρωί, ξέρετε, έχουμε και εκλογές για τους αντιπροέδρους. 9 το πρωί αύριο. Γι' αυτό παρακαλώ τους συναδέλφους, εφόσον επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, να είναι παρόντες στις 9 ακριβώς αύριο. Θα το επαναλάβω και πάλι. Πρέπει να τηρηθεί σήμερα το χρονοδιάγραμμα. Και έτσι περνώ στις ανακοινώσεις του Προέδρου, που δεν υπάρχουν. Σημείο 3. Αξιολόγηση της υλοποίησης προγράμματος ορίζοντας 2020 με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή της και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο. Ο κύριος Τόρβαλτς είναι ο εισηγητής. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ιδιαίτερη ικανοποίηση. Να μπορώ να παρουσιάσω το όριζον 2020 ως εισηγητή στην Επιτροπή των Προπολογισμών. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα με σαφή προσθεμένη αξία. Ξέρετε ότι υπάρχουν στατιστικέ για το κάθε ευρώ που δαπανάτε, για την έρευνα και την καινοτομία, που παράγει το 1 ευρώ 11 ευρώ άμεσα ή έμεσα οικονομικά ωφέλη χάρη στην καινοτομία, τις νέες εφευρέσεις, τα νέα προϊόντα. Το ποσοστό επιτυχίας στον το 2020 δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό, τόσο καλό όσο αυτό των προκατόχων προγραμμάτων για διάφορους λόγους. Πρώτον, επικαλύψεις καθώς οι διαδικασίες είναι διαφορετικές από τις στο παρελθόν. υπολογίζονται και οι εγκεκριμένε αιτήσει και οι νέε. Και αυτό σημαίνει διπλή δουλειά. Δεύτερον, το ενδιαφέρον ε, για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, αυξηθεί καθώς έχουν μειωθεί οι εθνικοί προϋπολογισμοί για το ίδιο θέμα. Ελπίζω ότι η Επιτροπή Ήτρα και η Επιτροπή θα εστιαστούν κυρίως στο δεύτερο τμήμα. Εγώ θα μιλήσω για το πρώτο. Εμείς το δεύτερο έχουμε να συζητήσουμε τα θέματα του προπολογισμού. Η στρατηγική λοιπόν ε, για το 2020 λέει ότι θα πρέπει να τίνουμε στο 3% επί του ΑΕΠ για την έρευνα και την καινοτομία. Πρόκειται για κοινό στόχο και για το εθνικό, αλλά και για τα, για τα εθνικά, αλλά και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά με περικοπές στους εθνικούς προπολογισμού, το ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να ενισχύσει τη χρηματοδότηση για την επιτεύξη των στόχων, κάτι βεβαίω το οποίο δύσκολα επιτυγχάνεται σε έναν προπολογισμό συμπιεσμένο από διάφορες πλευρέ. Αυτό ισχύει και για το προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο μετά τον ορίζοντα 2020. Γιατί θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τη χρηματοδότηση. Λόγω του περιορισμού σε τυπογραφικούς χαρακτήρες έχουμε παραλείψει αναφορές στο έτσι στη γνωμοδότηση. Ξέρουμε όμως ότι είναι οι περικοπές αυτές σημαντικές, πρέπει να κάνουμε τοπολογίες και εγώ προσωπικώς. Επίσης μια αναφορά στο Brexit καθώς ακόμα δεν έχει γίνει επίκληση από το Ηνωμένο Βασίλειο του άρθρου 50, αναμένεται όμως για την επόμενη εβδομάδα, δεν περιλαμβάνεται. Στον ορίζοντα πάντως θα έχουμε σημαντικό, σημαντικές συνέπειες από τις προσεχείς διαπραγματεύσεις για το Brexit, το οποίο θα επηρεάσει άλλωστε, οι οποίες διαπραγματεύσεις άλλωστε θα επηρεάσουν και το προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο με περικοπές 1% επί του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου που θα έχει βγει, επομένω θα είναι ακόμα λιγότερα τα χρήματα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αν υπάρχουν τώρα διαφορετικέ δυνατότητε ε, για την έρευνα και τεχνολογία, ώστε να διατηρηθούν τα επίπεδα τη χρηματοδότηση, ε, η δραστηριότητα ή αν ε, θα παραμείνει στο προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο, η έρευνα και η τεχνολογία, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Όπως είχε πει ο κύριος Ράμσφελτ μετά το 2001, υπάρχουν known unknowns, γνωστά, ε, γνωστοί αστάθμητοι, και unknown unknowns, άγνωστοι αστάθμητοι παράγοντες, όπως είχε πει ο κύριος Ράμσφελτ. Λοιπόν, χρόνο πολύ δεν έχουμε. Προς το παρόν αυτά έχω να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συντάκτη. Και τώρα καλώ τους συναδέλφους να λάβουν το λόγο. Χώσε Μανώλη Φερνάνδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να συμφωνήσω συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο συνάδελφος Τόρβαλτ. Ο στόχος που είχαμε ως πρώτη στρατηγική Ευρώπη 2020, το 3% του ΑΕΠ για την έρευνα και την κοινοτομία. Αυτά θα πρέπει να είναι μια προσπάθεια όχι μόνο του δημόσιου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού. Οι επιχειρήσει θα πρέπει να κάνουν την προσπάθεια για αυτέ οι ίδιε. Και βεβαίω τα διευθυντικά ταμεία θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Υπάρχουν πολλές συμφωνίε εταιρικής σχέσης, όπως στην Πορτογαλία, που λαμβάνουμε όσο μπορούμε υπόψη τη διάσταση τη έρευνα και κοινοτομία. Όμω, είναι γεγονό ότι ορίζοντα 2020 και των 500 εκατομμυρίων ευρώ είναι ένα ποσό σημαντικό για την ε, ανάπτυξη στην Ευρώπη και την πρόοδο της έρευνας και κοινοτομίας. Βλέπουμε πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα και δύο κουβέντες γιατί ο Επίτροπος έχει κάνει ε, πολύ σημαντική δουλειά στο θέμα αυτό και θα πρέπει να δούμε και τον, ε, το πόσο μπορεί να ανοίξει ο ορίζοντας 2020 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα εργαλείο σημαντικό, καθοριστικό να μην ξεχνάμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά τη ευρωπαϊκή οικονομία σε μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα πρέπει λοιπόν ο ορίζοντα 2020 να μα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε και πολλά τα κοινωνικά προβλήματα και δυσκολίε και προ την αύξηση του πληθυσμού. Ε, το θέμα τη ε, συμπερίληψη και τη ένταξη, τη κοινωνική ε, συνοχή. Είναι θέματα σημαντικά όπου ο ορίζοντα 2020 μπορεί να προσφέρει με την παρουσία του. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν το στηρίζουμε και θα πρέπει να συμπληρώνεται όχι μόνο από τα διευθυντικά ταμεία και τα κονδύλα για την έρευνα που διαχειρίζονται τα κάτι μελη αλλά και με προγράμματα που θα ασχολούνται με την ένταξη και τις κοινωνικές προεκτάσεις. Το ίδιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο των Στατικών Επενδύσεων, το γνωστό ως πρόγραμμα Juncker, το ΕΨΙ, και εκεί είναι σημαντικό να δούμε τις δυνατότητες ε, συμπληρωματικότητας και συνεργασίας έχει φανεί ότι και το ΕΦΣΥ μπορεί να συνεισφέρει ώστε ορίζοντας 2020 επιδιώκει σωστά τους στόχους του. Έρευνα και καινοτομία. Και ότι εξυπηρετεί και την οικονομία και τους ίδιους τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έιντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος ε, της ε, σκιώδους ε, εισηγητρίας από την ομάδα μου της Κλέρ Μούντι που δεν μπορούσε να έρθει. Εξ ονόματος της όμως θα κάνω εγώ κάποια σχόλια. Το πρώτο είναι, θέλω να ευχαριστήσω για την γνωμοδότηση των συναδελφών Ε, Συμφωνούμε σε αντρές γραμμές με τις ιδέες που επισημαίνει. Θεωρούμε ότι ορίζον 2020 είναι ένα πρόγραμμα που προσέχτηκε ιδιαίτερα στην Επιτροπή Προπολογισμών είδαμε, παρακολουθήσαμε την εκτέλεση του προγράμματος και από δημοσιονομικής πλευράς αλλά και επί της ουσίας, ό,τι αφορά δηλαδή την επίτευξη των στόχων που είχαμε θέσει. Βέβαια εμείς εστιάζουμε εδώ πιο πολύ στη χρηματοδότηση. Συμφωνούμε με αρκετές από τις προτάσεις του κυρίου Τόρβαλς για τη βελτίωση του προγράμματος Horizon 2020. Θεωρούμε επίσης σημαντικό να τονίσουμε ιδίως τον αρχικό στόχο του προγράμματος Ορίζω 2020 που έχει να κάνει με την επιστημονική αριστεία. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην ομοδότηση. Επίσης, σημαντικό θεωρούμε ε, να δοθεί προσοχή στην πρόταση της Κομισιόν για το European Innovation Council και πώς αυτό θα επιδράσει με το European Research Council και το COSME. Αυτά τα τρία προγράμματα επίσης. Πώς θα επηρεάσουν τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, το είπαμε βέβαια και ξανά και ξανά στην Επιτροπή μας, ιδίω δε όταν συζητούσαμε τη χρηματοδότηση του ΕΦΣΙ στην Επιτροπή μας, ασκήσαμε έντονη κριτική και προσπαθήσαμε να τροποποιήσουμε την πρόταση σε ό,τι αφορά το κατά πόσο θα έπρεπε να βγουν κονδύλια από το ορίζοντα 2020 για να χρηματοδοτηθεί το ΕΣ. Ξέρετε ότι μια από τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας σε όλες τις οικονομικές χρήσεις είναι λίγο-λίγο να ε, επιστραφούν αυτά τα χρήματα, αυτά τα κονδύλια που αφαιρέθηκαν τον του 2020. Θεωρούσαμε ότι ήταν σφάλμα αυτό που έγινε αρχικά, δηλαδή να αφαιρεθούν κονδύλια από ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο την, ε, την ε, επιστημονική αριστεία και να δοθούν αυτά τα κονδύλια στο ΕΦΣΙ. Μπορεί να δοθούν τα χρήματα σε παρόμοιου τομεί, ωστόσο το είδο δραμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται με τον ορίζοντα 2020 δεν είναι τα ίδια με αυτά που θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ. Τέλο πάντων, με αυτέ τι αποχρώσει ε, πρέπει να πω ότι συμφωνούμε με την πρόταση του κυρίου Τόρβαλ. Uh, Ευχαριστώ, Έντερ. Θα ήθελε κάποιο άλλο να πάρει το λόγο. αν όχι να ξαναδώσω το λόγο στον γιατί εφόσον θέλει να προβεί σε συμπληρωματικά σχόλια. Κύριε Στόρβαλ, σε ευχαριστώ, θα είμαι σύντομο. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα σχέδια για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Εγώ μελετούσα και την ιστοσελίδα της Κομισιόν ε, για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο και βλέπω ε, ότι κάποιες εξελίξεις υπάρχουν. Βέβαια ήταν πολύ διάσπαρτες οι πληροφορίες, ε, κάτι κατάλαβα, αλλά το πρόβλημα το βασικό είναι το τι θα γίνει με τον προπολογισμό, άπαξ και βγει εκτό το Ηνωμένο Βασίλειο και ταυτόχρονα έχουμε και τα δορυφορικά και κάπως είναι στριμωγμένα τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολύ στενά δημοσιονομικά περιθώρια με το Brexit είπε και ο Χωσέ Μανουέλ, είπε και η Έντερ. Νομίζω ότι συμφωνούμε με ό,τι αφορά τις ΜΜΕ, την αριστεία και όλα αυτά τα οποία θέλουμε να επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Rapporteur. Um, seems we have consensus here in the room that Horizon 2020 is ναι, έχετε δίκιο γιατί το ορίζοντα 2020 έχει μια πολύ σημαντική λειτουργία για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα δούμε ε, ώστε να υπάρξει και ένα κληροδότημα για την επόμενη θητεία και σίγουρα θα επηρεαστεί και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο στο σχεδιασμό του. Εκεί θα χρειαστεί να ρίξουμε άλλη μία ματιά για να βεβαιωθούμε για την προστιθέμενη αξία που επιδιώκουμε και ότι επιτυγχάνουμε τι νέε προτεραιότητε. Ο ορίζοντα 2020 θεωρώ ότι είναι το κλειδί για να δημιουργηθούν θέσει εργασία, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Προσωπική παρατήρηση θα έλεγα ότι το ορίζοντα 2020 είναι άκρο σημαντικό και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Τελείως προσωπική παρατήρηση, αλλά ελπίζω ότι σε δύο-τρία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετέχουμε ακόμη πλήρως και ότι θα συνεισφέρουμε προ του στόχου του ορίζοντα 2020. Οπότε μερικά από αυτά που είπατε μπορεί και να μην συμβούν, ελπίζω. Ε, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σα. Να σα θυμίσω ότι Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει 23 Μαρτίου λήξη για την, υποβολή, για την προθεσμία της υποβολής των στη μία το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 25 Απριλίου και στην Ήτρε, που είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, στις 29 Μαΐου. Ευχαριστώ. Σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2018. Τμήμα 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο λόγος των εισαγητή που είμαι εγώ ίδιος. Θα ήθελα να κάνω ένα-δυο σχόλια, συνάδελφοι. Ήδη έχουμε οργανώσει αρκετέ συναντήσει με του κέντρου τους Του ευχαριστώ για τι συνεισφορέ του. Είχαμε κάποιε επικοδομητικέ ε, συζητήσει ω τώρα. Και θα συναντηθούμε στη συνέχεια με τους δύο αντιπροέδρους του Προεδρείου στις 6.30 το βράδυ σήμερα. Ε, με κάποια έκπληξη πρέπει να σημειώσω στους συναδέλφους της Επιτροπής ότι Κανείς από την Επιτροπή μας δεν ε, παρέστην στις συνεδρίες του Προεδρείου που ε, αναμενόταν να συζητηθούν οι προτάσεις ε, αυτής της πρότασης. Αυτό κάπως με ευνηδίασε και επίσης με ευνηδίασε που η διάσκεψη των Προέδρων έλαβε την απόφαση να με γίνει συζήτηση για το θέμα στην Ολομέλεια για τις εκτιμήσεις που αφορούν τον προβολισμό του Κοινοβουλίου. Εδώ λοιπόν να σας αναγγείλω ότι αυτό που προκύπτει από τη συνεδριάση των σκιωδών είναι ότι υπάρχει στήριξη γενικώ από την Επιτροπή μας. Υπάρχει αποφασιστικότητα για το επίπεδο, μάλλον υπάρχει μια απόφαση για το επίπεδο των δαπανών. Μια απόφαση να ακολουθήσουμε την παράδοση της Επιτροπής μας. Οι δαπάνες να είναι κάτω του 20% του τίτλου 5 και ο στόχος που συμφωνήσαμε να έχουμε είναι ότι ό,τι αύξηση υπάρξει να μην ξεπεράσει το επίπεδο του πληθωρισμού. 1,7%. Από ό,τι φαίνεται η πρόταση που έχουμε είναι στα, πρώτα, στα στάδια βέβαια ακόμα, αλλά η, πρώτα, αύξηση είναι 0,95%. Τα θέματα που έχουν συζητηθεί περισσότερο στο επίπεδο αυτού του πληθωρισμού είναι το θέμα των κτηρίων με ιδιαίτερη μέρημνα για το PHS ή η ασφάλεια τις εκλογές του 2019 και την προκυλοκή εκστρατεία που θα χρηματοδοτηθεί εκ των προτέρων, κάποια από αυτά τα κονδύλια θα δαπανηθούν ήδη το 2018, και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών βιβλιοθήκης. Αυτά είναι τα θέματα σε σημεία. Οι σκιώδες τα γνωρίζουν, τα έχουμε συζητήσει και γνωρίζουν, ελπίζω επίσης, ότι θα συνδεθούμε στις 6.30 για την πρώτη συνδιαλλαγή. Έχουμε επίσης λάβει 204 τροπολογίες για την αρχική έκθεση, τις οποίες αυτή τη στιγμή μελετούμε και επεξεργαζόμαστε. Ευχαριστώ όλες και όλους όσους και όσους υπέβαλαν τροπολογία. Και ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τις πολιτικές ομάδες με τη σειρά. Ο Χώζε Μανουέλ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω δίνοντα έμφαση στο ότι εξήρετε συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε και την ποιότητα με την οποία φέρνετε ει πέρα στο όλο θέμα, την έκθεση και του στόχου τη. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προπολογισμό επενδύσεων. 94% αφορούν την ε, τις επενδύσεις και το 6% αφορούν τις δαπάνες όλων των θεσμικών οργάνων. σε αυτό το 6% του ευρωπαϊκού προπολογισμού, ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου, με συγχωρείτε, ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου επίση ανέκαθεν δεχόταν επιθέσεις και επικρίσεις. Όταν ο στόχος που πρέπει να έχουμε, ο πρωταρχικός, είναι της α, ε, κοινοβουλευτικής αριστείας και δεν επιτυγχάνεται, υποτίθεται. Δηλαδή, υπάρχει νομοθεσία χωρίς ε, την κατάλληλη ποιότητα. Αυτό ε, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όταν η νομοθεσία θεωρείται κακή υπάρχει και κόστος για τους πολίτες. Εδώ λοιπόν έχουμε εξαιρετικούς συνεργάτες, εξαιρετικούς ε, συμβούλους των πολιτικών ομάδων, συνεργάτες από τη γραμματεία που εργάζεται πολύ αποτελεσματικά, πολύ καλή ποιότητα στην ερμηνεία και τη μετάφραση όλων αυτών ε, των στοιχείων που αφορούν. 94% επενδύσεις και 6% για όλα τα θεσμικά όργανα, για όλες τις διοικητικές δαπάνες. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής μας έχει κάποιο παράδειγμα ανάλογα από τη χώρα του, το Ηνωμένο Βασίλειο, κάποιο έστω δημόσιο φορέα, όπου μόνο το 6% να καλύπτει τι δαπάνε. Τι δαπάνε του διοικητικού προσωπικού. Δεν νομίζω να έχετε κάτι τέτοιο να μας παραθέσετε. Εγώ δεν γνωρίζω κανένα θεσμικό όργανο όπου μόνον το 6% αφιερώνεται στις διοικητικές δαπάνες. Τέλος πάντων, η ερμηνεία που συνήθως δίνεται 6% το επαναλαμβάνω για όλα τα θεσμικά όργανα. Την Επιτροπή των Περιφερειών, την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή, τον Επιτροπή του Συμβούλιο, Και από αυτό το 6% χρησιμοποιείται λιγότερο από το 20% ε, από το Κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε κυρίω του στόχου του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και πώ θα επικοινωνούμε καλύτερα, πώ θα προβάλλουμε καλύτερα όλα αυτά προ του Ευρωπαίου πολίτε. Θέλουμε να συμμετέχουν περισσότερο στι εκλογέ και αυτό να γίνει ήδη από το 2019. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν μια προεκλογική εκστατεία για να ενημερωθούν για όσα κάνουμε, αλλά και να πληροφορηθούν, να ενθαρρυνθούν, να πάρουν κίνητρα για να συμμετέχουν περισσότερο οι νέοι ψηφοφόροι. Όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την ασφάλεια των κτηρίων και την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων, των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Εδώ λοιπόν Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο προπολογισμό δεν μπορεί να είναι μηδενικό. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που δεν προ την ολοκλήρωση τη εκτέλεσή του, όπω στα κτίρια ή στι ανακαινήσει. Αλλά ο προπολογισμό πρέπει να εξασφαλίζει κάποια συνέχεια. Και όταν μιλάμε για συνέχεια, χρειάζονται και συμβαστικέ λύσει είτε στα, ε, στο επίπεδο των κτηρίων, της ανακαίνησης, είτε των θεμάτων των ε, βουλευτών, δεν μπορεί να ξανανοίγουν όλες αυτές οι κουβέντες σε κάθε διαδικασία προπολογισμού. Γιατί πάντοτε ξεκινάει μια συζήτηση για τα θέματα αυτά που οδηγούν τελικά πρώτα σε συζήτηση και μετά σε λαϊκιστικές παρεκτροπές. Πρέπει λοιπόν εδώ να είμαστε σαφεί στην γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε, να προβάλλουμε σωστά το έργο μας ε, στι επίσημε γλώσσες τη Ένωση. και επίσης πρέπει να έχουμε ένα θεσμικό όργανο αποτελεσματικό από όλε τι ε, οπτικέ γωνίες και την περιβαλλοντική ακόμη. Είναι και αυτό σημαντικό. Πρέπει η αποτελεσματικότητά μα να είναι και να διαφαίνεται σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και σε αυτό των δαπανών. Πρέπει να επιζητήσουμε την κοινοβουλευτική αριστεία ως στόχο χρησιμοποιώντας όσο λιγότερους πόρους γίνεται. Αυτό όμως το ελάχιστο των πόρων σημαίνει ότι χρειάζονται και οικονομικοί πόροι για να επιδιωθεί ο στόχος της κοινοβουλευτικής αριστείας. Οπότε, δαπάνες θα υπάρχουν. Υπάρχουν ε, αυτές οι δαπάνες που πρέπει να γίνουν, πρέπει να εκτελεστούν και βεβαίως Εφόσον αυτές οι αρχές διαδικηδεύονται, θα πρέπει να, ε, να κάνουμε και τις περικοπές μας, να κάνουμε οικονομίες όσο μπορούμε, αλλά μην ξεπεράσουμε και το όριο του λογικού. Μην βλάψουμε τα ίδια τα συμφέροντα των πολιτών με τις περικοπές. Αυτό είναι ο στόχος της δουλειάς μας. είναι βέβαιο ότι θα πετύχουμε κάποια συμφωνία και καθώς θα πλησιάζουμε προς το τέλος της θητείας διαρκώς θα προκύπτουν αυτοί που θα χρησιμοποιούν τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου ως πρόσχημα για να κάνουν εκστρατεία κατά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ακόμα και οι ίδιοι αυτοί που λαμβάνουν χρήματα από τον προπολογισμό της Ένωσης για να πάρουν αφορμή και να επιτεθούν να ταπεινώσουν, να υποβαθμίσουν τις γυναίκες. Άλλοι που παίρνουν λεφτά από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για να επιτεθούν και να αμφισβητήσουν την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και την Ένωση. Αυτά όμως είναι όσα συμβαίνουν ε, σε ένα κοινοβουλευτικό σώμα και πρέπει να σεβαστούμε και την αρχή της αντιπροσώπευσης των πολιτών. Απλώς δεν μπορούμε και να ενδώσουμε στις ε, ακραίες και ριζοσπαστικές τοποθετήσεις, είτε είναι της ε, δεξιάς είτε της αριστεράς, που όλο ένα αναδύονται και πιο ισχυρές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει μικρόφωνο δυστυχώ ο μιλητή και δεν τον ακούμε. Okay, thank ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρά τη δουλειά που ο Πρόεδρος και συγκεκριτής μας ε, έχει φέρει σπέρας, με τις 204 τροπολογίες που πρέπει να μελετηθούν, αρκετή δουλειά, και προφανώς έχει προκαλέσει και συζητήσει η όλη έκθεση, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτή τη φάση. Δεν θα περάσω στο σχόλια των λεπτομεριών. Η συνδιαλλαγή, όπως είπατε, αρχίζει έτσι και αλλιώς απόψε. Πρέπει να κάνουμε επαφές με τις ομάδες μας, με τον εισηγητή, με τους συνεργάτες των ομάδων. Θα ήθελα λοιπόν όπω έκανε ο συνάδελφο και φίλο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντε, να κάνω κάποιε γενικότερε παρατηρήσει. Και θα ξεκινήσω ευχαριστώντα τον συγκεκριτή για τη δουλειά του, είναι εξαιρετική. Και να μην ξεχνάμε και το πλαίσιο εντό του οποίου διεξάγονται αυτέ οι διαπραγματεύσει. Ε, έχουμε συναντήσει των σκιωδών, διμερεί επαφέ διαρκώ. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει βούληση να γίνει μια καλή λογική δουλειά. Βεβαίω υπάρχουν κάποια σημεία αναφοράς. Αναφέρθηκαν αυτά. Ε, η αύξηση των ε, δαπανών δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό του πληθωρισμού. Αναφέρθηκε αυτό. Είναι και λογικό. Και η δική μου ομάδα έχει κάνει σχετικέ προτάσει για την επιδίωξη του στόχου αυτού. Αλλά υπάρχει μια σημαντική δουλειά να γίνει για να μην ε, έχουμε προβλήματα ως προς την αποτελεσματικότητα και να γίνουν όλα αυτά στα πλαίσια της λογικής. Η δική μου η μελέτη των προβλημάτων του προπολογισμού ε, με τα οποία έχω σχοληθεί πολλές φορές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι θέματα που τα έχω σχολιάσει και στις συναντήσεις των σκιωδών. Υπάρχουν οι εξή αρχές. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε την αρχή της διαφάνειας. Θα πρέπει οι πολίτες και όλοι να γνωρίζουν τι δαπανάτε, πώς και πώς ασκείται ο δημοκρατικός έλεγχος. Αυτό είναι μια αρχή από την οποία δεν μπορούμε να, από την οποία δεν μπορούμε να τρεπόμαστε. Ε, επίσης η αποτελεσματικότητα. Πρέπει έστω και το τελευταίο λεπτό του ευρώ που χρησιμοποιείται να ξέρουμε ότι συνεισφέρει στην εκπόνηση της σωστή ε, νομοθεσίας και το καθεξής. Και υπάρχει και μια αρχή που πρέπει να ακολουθήσουμε, μια αρχή αρνητική, η καταπολέμηση ε, των ε, ατασταλιών. Υπάρχουν πολλές απαιτήσει από τους πολίτες, πολλές απαιτήσει από τους πολίτες, όχι λαϊκιστικής προέλευσης, λαϊκής θα έλεγα, που εκμεταλλεύονται τον προπολογισμό για να επιτεθούν στην ε, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, στο ίδιο το λειτουργήμα του βουλευτού με αφορμή τον προπολογισμό. Εδώ λοιπόν πρέπει οι αρχές, να γίνονται, οι αρχές αυτές να γίνονται σεβαστές σε όλους τους τίτλους και σε όλα τα κεφάλαια του προπολογισμού. Υπάρχουν πολλά θέματα λοιπόν ε, με τις ε, περικοπές και τις προσαρμογές που θα μπορούσαν να γίνουν για παράδειγμα, η ομάδα μου προτείνει τις γραμμές του προπολογισμού που διαρκώς ε, υπερτιμούνταν. Κάποια ποσά πολλές φορές παραμένουν αδαπάνητα και μετά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, για άλλους σκοπούς. Ας τα προσαρμόσουμε από τώρα. Ή η αρχή που μόλις ανέφερα, η αρχή της αποτελεσματικότητας. Πρέπει να γίνεται σεβαστή, είναι θεμελιώδης. Πρέπει να δούμε τους τίτλους των ε, κονδυλίων που είναι άκρος απαραίτητα. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς, σαφείς στους στόχους των ε, κονδυλίων, δηλαδή για τους οποίους θα, εκτελ, εκτελούνται τα ποσά αυτά. Και να είμαστε βεβαίοι ότι υπάρχει η accountability, η λογοδοσία σε σχέση με τη δαπάνη αυτών των ε, ποσών. Αυτή ήταν η κατευθύνια γραμμή, η Τη παρέμβασή μου και τη συλλογιστική μου, τη δική μου και τη ομάδα μου. Αυτό που θα μπορούσε να προκύψει είναι τα βασικά κόμματα του Κοινοβουλίου να φροντίσουμε να συνασπιστούμε για το θέμα αυτό, να πετύχουμε μια κοινή θέση για να αξιοποιήσουμε στο δυνατόν περισσότερο τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και να στηρίξουμε την ε, ευρωπαϊκή πορεία, την πορεία της Ένωσης. Η δική μου η ομάδα δεν έχει καμία ελακιστική δημαγωγική διάθεση και θα παραμείνει στο πλευρό αυτών που θα επιδιώξουν την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Thank you. Uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν ε, θα ξαφνιάσω κανέναν, φαντάζομαι, ευχαριστώντας θερμά τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά του. Σας ευχαριστώ κύριε Κερμέλ. Εδώ ε, έχουμε δει πολλά πράγματα, έχει περιλάβει στην εγγραμματευσή του πράγματα που δεν είναι καθόλου απλά ή αυτονόητα. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια των ε, προαλεξάντων, αλλά σε ορισμένα διαφωνώ. Έχω την εντύπωση ότι εδώ ανοίγουμε ένα μέτωπο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ένα μέτωπο δηλαδή εκείνων που, λέει, που λένε ότι θα πρέπει να δαπανούμε περισσότερα, ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες δαπάνες, ότι πρέπει να ε, δίνουμε πολλά χρήματα για το κοινοβούλιο και εκείνων που λένε θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιες οικονομίες ε, στις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όποιος το λέει αυτό φαίνεται σαν να είναι εχθρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θέλει να βλάψει την αποδοτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν ε, λάθος άλλωστε και παραπλανητικό να κάνουμε συσχετισμούς με τον τρόπο λειτουργία άλλων, των εθνικών δηλαδή κοινοβουλίων, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δική του δομή, ε, ιδιάζουσα. Δεν ελέγχουμε καμία κυβέρνηση ή κυβερνητικό μηχανισμό. Έχουμε δικό μας τρόπο λειτουργίας και γι' αυτό τέτοιου είδου παραλληλισμοί δεν βοηθούν. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να πράξουμε αυτό το οποίο πράττουμε. Συνήθως να, να κοιτούμε εάν τα χρήματα που έχουν ταπανηθεί εξυπηρέτησαν το στόχο για τον οποίο είχαν προβλεφθεί και εάν εξυπηρετούνται οι στόχοι μας. Και σε αυτό μπορούμε να είμαστε περήφανοι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι η αποδοτικότητα, κατά την άποψή μου, της χρήσης του προπολογισμού είναι υψηλή. Πρέπει να διατηρηθεί υψηλή. Μπορεί να βελτιωθεί ασφαλώ και οφείλουμε να το πράξουμε αυτό, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να θεωρεί κανεί ότι είναι ιερά και όσοι ορισμένα κεφάλαια του προπολογισμού και ότι μπορούν να γίνουν περικοπέ ή εξοικονομήσει πόρων πουθενά. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ. Κύριο Δεπρέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα και στο παρελθόν την ευκαιρία να εκφράσω την εκτίμησή μου για την έκθεσή σας στις γενικές γραμμές της, τουλάχιστον στο γραπτό κείμενο, στο φιλολογικό θα έλεγα τμήμα. Α, σε σχέση με τα αριθμητικά όμως ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, λέτε και ελπίζω να κατάλαβα εγώ λάθος, ότι θέλατε τον περιορισμό του προϋπολογισμού, την αύξηση του προϋπολογισμού για το 2018 να την περιορίσετε στο 0,95%. Ελπίζω να να παρεξήγησα εγώ τα λόγια σας. Και γιατί. Γιατί αν λάβουμε υπόψη το 68% των ταπανών του Κοινοβουλίου είναι σχετικές με το προσωπικό. Ότι έχουμε πολύ περιορισμένο περιθώριο κινητικότητα σε σχέση με τον υπολογισμό του συστήματος τη τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που είναι προσδιορισμένο σύστημα αυτό το 68% μπορεί να οδηγήσει σε 3,0 ή 3,2% αύξηση. Εάν λοιπόν ε, επιμένετε για 0,95% αύξηση σε, σε πολλά κεφάλαια θα πρέπει να κάνετε περικοπές, λαμβανομένου υπόψη του θέματος της θυμαριθμικής ε, αναπροσαρμογής. Και σε σχέση με τον προπολογισμό του 2015 πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε χαμηλότερα επίπεδα Άρα δεν μου φαίνεται εφικτό τεχνικά αυτό που προτείνεται. Έχω λοιπόν τις επιφυλάξεις μου και επίσης δεν θυμούμε η Επιτροπή μας να έχει συμφωνήσει σε τέτοιου είδους ποσοστά. Ούτε καν στη συνάντηση των συντονιστών και γίνεται τη συζήτηση, τέτοια τι απόφαση. Δεύτερον, σε σχέση με το ύψος των ε, εξοικονομήσεων πόρων, είχα ορίσει έναν ε, κανόνα και τον επιβεώνω σήμερα, ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, οικονομία να κάνουμε στις δημοσιονομικές εκείνες, ε, στα δημοσιονομικά εκείνα κονδύλια, στα οποία έγινε ανάκτηση στο πλαίσιο του ραμασάζ κονδυλίων τα τελευταία τρία χρόνια συνεχώς. Αλλά γι' αυτό και εδώ απευθύνομαι στην γραμματεία του Κοινοβουλίου, στη διοίκηση, του Γενικό Γραμματέα δηλαδή και τη διεύθυνση ΦΙΝ, πρέπει να έχουμε ακριβή στοιχεία. Γιατί τα στοιχεία που μας δώσατε δεν είναι σαφή. Αφενός μεν μας λέγεται ότι για να χρηματοδοτηθεί το πλαίσιο στο τρέχουσα χρονιά χρειαζόμαστε 60 εκατομμύρια περίπου. Εγώ βλέπω ήδη 32 εκατομμύρια πρόβλεψη. Τα 32 εκατομμύρια μας λέτε όμως δεν είναι μέρος αυτών των 62 εκατομμυρίων. Εξηγήστε μας λοιπόν τελικά τι έχετε προβλέψει για τον προϋπολογισμό τώρα, για τη χρηματοδότηση του πλαισίου και δεν μιλώ για τα λοιπά, ε, παρελκόμενες δαπάνες για μικρό επιδιορθώσεις και τα λοιπά. Πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα γιατί δεν είχαμε ποτέ το θάρρος και αυτό είναι κοινή δηλία θα έλεγα να μιλήσουμε ανοιχτά για το πλαίσιο της χρηματοδότησης των κτηρίων και ιδίω του ΚΑΔ ε, και πάντοτε αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του ραμασάζ. Ας ε, κοιτάξουμε λοιπόν πόσα πρέπει να, προβλέψουμε για τη χρηματοδότηση του ΚΑΝΤ, ώστε να μην αναγκαζόμαστε πάντα να προσφεύγουμε σε αυτή τη λύση των υπόλοιπων ε, ποσών. Αυτό το αίτημα λοιπόν προς το Γενικό Γραμματέα και την Γενική Διεύθυνση των Οικονομικών. Επίσης, και μια... κύριε Πρόεδρε και κύριε Ισηγητά, έχετε διπλό ρόλο σήμερα, δεν βλέπω πως σε ορισμένα σημεία ξεπερνάτε τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα. Σε ορισμένε ε, γραμμέ του προπολογισμού, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ γενναιόδωρο ο Γενικό Γραμματέα και σα βρίσκω ακόμη πιο γενναιόδωρο. Μήπω υπάρχουν κάποιε εκφράσει αλληλεγγύη που μου είναι άγνωστε ή κάποιοι λόγοι που δεν ε, μου είναι εκεί. Πάντως σε κάποιες άλλες γραμμές, πολύ σημαντικές και πολιτικά ευαίσθητες, προβαίνεται σε ε, περικοπές που θέλετε να φτάσουν ε, έως το 2016 μόνο, για να μην πάνε στο 2017. Μα γιατί αυτό, αφού είχε προβλεφθεί ότι θα πάρει μέχρι το 2017, γιατί να ε, μην ε, τις αφήσουμε έτσι και να θέλουμε να τις περιορίσουμε στο 2016. Τελευταίο στοιχείο. Πρέπει να γίνει μια πραγματική συζήτηση για τα εκατομμύρια που προβλέπονται ειδικά για την επικοινωνιακή πολιτική που αφορά την, ε, το πρόδρομο, θα έλεγα, της προεκλογικής εκστρατείας. Και διαρωτώ με ώρες ώρες εάν ε, η Διεύθυνση για την Επικοινωνιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει λάβει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι, όπως ξέρετε, ε, χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα κοινωνικά δίκτυα, η επικοινωνιακή πολιτική προς τους νέους, σε αυτό πρέπει να στηρίζεται. Ενώ βλέπουμε ότι ακόμη χρησιμοποιείται το έντυπο, ή άλλοι τύποι επικοινωνίας. Επίσης βλέπω πολύ χρήμα να διοχετεύεται στα κτίρια. Τι θα τα κάνουμε τα κτίρια στις εποχές της νέας τεχνολογίας και της τεχνολογίας. Υπάρχουν γραφεία επικοινωνιακής ε, πολιτικής ή ενημέρωσης καλύτερα. Ποιος θα πάει εκεί. Ε, μόνο ο ακριβή υποστηρικτής ή τελικά κάποιος ο οποίος θα μπορούσε και παλού να αντλήσει τις πληροφορίες. Ας ε, επανεξετάσουμε λοιπόν τη στρατηγική επενδύσεων στα κτίρια, ας επανεξετάσουμε τη στρατηγική των επενδύσεων στο έντυπο και ας βρούμε λύσεις άλλες γιατί στη στρατηγική της επικοινωνιακής ε, της επικοινωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βλέπω πραγματικά πουθενά επικοινωνία για το μέσο πολίτη. Πρέπει να είναι κανείς διανοούμενος για να καταλαβαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα οι, οι, οι λαϊκές τάξεις είναι αυτές οι οποίες τελικά ε, απομακρύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την απορρίπτουν. Ας απαιτήσουμε από τις ε, ε, υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτέλους να κάνει μια πρόταση για επικοινωνιακή πολιτική που θα στραφεί προς εκείνον στον οποίο δεν απευθυνόμαστε συνήθως και ο οποίος λέει «Μα δεν ξέρω τι είναι αυτοί, δεν ε, ταυτίζομαι μαζί τους, δεν καταλαβαίνω τι μου λένε αυτά τα θεσμικά όργανα». Συνοψίζοντα, δεν συμφωνώ με το 0,95% που προτείνατε. Πιστεύω ότι το επίπεδο των ε, περικοπών μπορεί να προσδιοριστεί μόνο όταν είναι γνωστό το πόσο θα χρειαστούμε για τη χρηματοδότηση του CAD του πρώην Adenauer, ε, του Adenauer για ε, τα μεταταραμασάζ. Επίσης ε, πρέπει ρητά να αλλάξει το σύστημα για να μην παίρνουμε τα για τη χρηματοδότηση του ΚΑΝΤ. Χρειάζεται μια στρατηγική ενημέρωσης επικοινωνιακή πριν να δεσμευθούν τα 25 εκατομμύρια και προσωπικός σας καλώ να με πείσετε για κάποιες δαπάνες που προτείνετε να αυξηθούν ενώ δεν βλέπω δικαιολογίες σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άσφορτ, ευχαριστώ πολύ. κύριος Ταράντ, παρακαλώ. Θέλετε το λόγο. δυστυχώ ναι, λέει ο κύριο Τάραντ. Ευχαριστώ πολύ. Για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια. Κάνατε καταπληκτική δουλειά. Και ηρωνικός πώς συγχαρητήρια που δεν εκλειφθήκατε σε μια σημαντική συνεδρίαση του Προεδρείου. Ο κ. Σαρτουή, από ό,τι θυμάμαι από πέρυσι, ναι, μεν είχε προσκληθεί, αλλά δεν το πετράπει είσοδο εγώ τα έχω συνηθίσει αυτά βέβαια γιατί γεννήθηκα στην ε, Σοβιετική Ένωση και υπήρχε αυτό το οι υψηλέ ε, συναντήσει όπου οι ε, κομμουνιστές η απλοί δεν μπορούσαν να συμμετέχουν. Ο κύριος Αρτουή όμως προέρχεται από την δημοκρατική χώρα που λέγεται Γαλλία και δεν είχε προσληφθεί. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι κι εσείς δεν χάσατε τίποτα. Λυπούμε που το λέω αυτό για τις διαδικασίες μας. Κάποιες σύντομες τώρα παρατηρήσεις σε σχέση με το τι ακόμη κατά την άποψή μου μπορεί να γίνει. Το πρώτο. Εκπηγάζει από την απόφαση της προηγούμενης χρονιάς για την δημιουργία 76 θέσεων για τις πολιτικές ομάδες. Βλέπουμε τώρα ότι αντισταθμίστε κατά κάποιο τρόπο με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα Βέλε με δημιουργία 50 τόσων θέσεων που τις πήραν βιαίως από την κοινοβουλευτική δομή και τις έβαλαν στις πολιτικές ομάδες. Τώρα βλέπουμε ότι πιο τίμιο θα ήταν να είχαν δοθεί απευθεία στι πολιτικέ ομάδε και να αναλυφθεί και η σχετική πολιτική ευθύνη για την απόφαση αυτή, κάτι το οποίο δεν έγινε. Αυτό νομίζω εννοούσε και ο κύριος Ντοσάντος αυτό σημαίνει ότι δίνουμε πειραμοχικά στους δημαγωγούς, στους λαϊκιστές ή αντιευρωπαίους, όπως άλλοι θέλουν να τους αποκαλούν, αντιευρωπαϊστές. Εγώ ενστικτοδός, αυθορμήτως ε, θα έλεγα ε, μην αντισταθμίσετε εκεί κύριε Γενική Γραμματέα. Μπορεί να είναι πιο δύσκολη επίτευξη αποτελεσμάτων όπως είπε και ο κύριος Φερνάντες. Στρέφομαι σε κάτι άλλο. Κατέθεσα ορισμένες τροπολογίες. 200 είπατε έχουν κατατεθεί, δικές μου είναι το 1%. Χαίρομαι. Πολύ σύντομα λοιπόν να, να κάνω κάποια σχόλια. Μπορεί να είναι λίγες, αλλά είναι σημαντικές αυτές οι τροπολογίες πιστεύω, διότι... Μιλάμε για τη βουλευτική επικουρία. Υπήρχε κάποια υπόσχεση που εκκρεμούσα αλλά δεν έγινε τίποτα. Κάναμε ένα μισό βήμα για αύξηση των αμοιβών των διαπιστευμένων συνεργατών, αλλά αναβλήθηκε εφαρμογή ο συνάδελφός μας, ο καλός συνάδελφος κύριος Ρούμπιχ, προτείνει να γίνει και το δεύτερο ε, μισό του βήματος, θες πάντων να καλυφθεί όλο αυτό, το, όλο αυτό, αυτή τη διαδρομή. Δεν ξέρω Υπάρχει μεγάλο συνασπισμό των μεγάλων ομάδων δεν υπάρχει. Ε, κατά την προσωπική μου άποψη όμω νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει, αν το επιτρέπει ο προπολογισμό με τα αυξημένα αυτά ποσοστά. Αλλά ακόμη και σε περίπτωση που δεν μπορούμε, θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες αδικίες. Μια εκ των οποίων είναι ότι πηγαίνουμε στο Στρασβούργο και εκεί οι απολαβές το προσωπικό είναι 40% υψηλότερη από αυτέ των διαπιστευμένων συνεργατών και αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ. Άνθρωποι είναι όλοι. Τρώνε το ίδιο, κοιμούνται στα ίδια ξενοδοχεία. Γιατί να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση λοιπόν του κόστου. Δεν το κατανοώ. Και ελπίζω να το πείτε στον Γενικό Γραμματέα ή σε οποιοδήποτε άλλο έχει λάβει αυτή την απόφαση ή λαμβάνει τέτοιε αποφάσει. Δεύτερον, Δεν θα εμβαθύνω σε αυτό, όμως νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια περαιτέρω ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Το τέλεφαξ βαρέθηκα πλέον. Είναι μια εφεύρεση Αμερικανική του 1969. Έλεος. Να τη χρησιμοποιούμε μεταξύ Βρεξελών και Λουξεμβούργου. Ε, μου δημιουργεί κάποιο άγχος. και νομίζω ότι ξέρουμε όλοι τι μπορούμε να κάνουμε. Email, μα δεν απαντούν στα email, γιατί σου λένε πρέπει να μας στείλετε με fax το κείμενο, το αντίγραφο. Και επειδή έρχομαι από μια απομακρυσμένη περιοχή, έχω ένα πρόβλημα με τις ομάδες επισκεπτών. Έχουμε τώρα ένα νέο, πολύ ωραίο σύστημα. Ουσιαστικά επιστροφή των εξόδων βασίζονται στις πραγματικές δαπάνες. Υπάρχουν όμως κάποια όρια. Και επειδή υπάρχει μονοπόλιο στις μεταφορές και άνθρωποι που έρχονται εδώ δεν είναι αυτάρκης, όπως πρέπει να άστεγοι, είχα καλέσει εγώ μια ομάδα αστέγων. Δεν δίνουμε παρκή χρηματοδότηση για αυτούς που ζουν ιδίως έστω μακριά από το κέντρο της Ευρώπης, στην περιφέρεια. Μια κάπως περίεργη παρατήρηση σε ό,τι αφορά την ε, εσωτερική ανάθεση των ε, υπηρεσιών ε, μεταφορών, τους οδηγούς. Είναι σημαντικό νομίζω να το ξέρει και ο συγητής. Σήμερα ρώτησα έναν οδηγό γιατί δεν χρησιμοποιεί ε, την, τον λεωφοριόδρομο για να παρακάμψει την κίνηση, όπως μπορούν να κάνουν κάποιοι οδηγοί κανονικοί και μου είπε ότι δεν μπορώ γιατί έχουμε εκμισθωμένα οχήματα προς το παρόν αλλά θα έχουμε σύντομα κοινοβουλευτικά. Επειδή είναι πιστός ε, υπηρέτης του κοινοβουλίου δεν μπορώ να αποκαλύψω το όνομά του. Αλλά υπάρχει τώρα ε, σχέδιο για αγορά νέων αυτοκινήτων, ενό νέου στόλου αυτοκινήτων. Υπάρχει πρόβλεψη στον προπολογισμό. Πώ θα το λύσουμε αυτό το ενδιαφέρον πρόβλημα. Και ξέρετε, κάποιοι οδηγοί δεν πήραν τη δουλειά διότι δεν μιλάγαν πολύ καλά αγγλικά. Εγώ δεν μιλάω γαλλικά. Το πρόβλημά μου είναι να βρει μια θέση ο οδηγός. Να βρει τη διεύθυνση. Συγγνώμη. <clears throat> Και όχι να έχουμε κουτσομπολιό μέσα στο αυτοκίνητο. Το θέμα να μπορεί να το δρόμο του άνθρωπος. Να έχετε υπόψη και αυτό λοιπόν. Και αυτό το αίμα που κάνει την ε, ύπαρξή μας πιο φιλοπεριβαλλοντική, μειώνει τα απόβλητα κτλ. Και υπάρχει βέβαια και μεγάλος ελέφαντας στην αίθουσα που είναι κτηριακή πολιτική, το είπαν και άλλοι. Πώς θα τον βγάλουμε από την αίθουσα ο ελέφαντας αυτός, είτε για το καντ, δεν θέλουμε άλλο ραμασάζ, είπε και ο κύριος Δεπρέ, ή για το Polar Respack που έχουμε έργα ανακαίνησης. πρέπει να κάνουμε την ερώτηση. Γιατί χρειάζονται αυτά τα χρήματα. Θέλουμε να μετακομίσει αυτός ο κόσμος από τα γραφεία του εκεί που θα γίνουν οι εργασίες, ενώ δεν ξέρουμε τι εργασίες θα γίνουν, γιατί ε, και πού χρειάζεται ανακαίνιση και πώς θα εκενώσουμε τους χώρους χωρίς να τα ξέρουμε όλα αυτά εκ των προτέρων. Αυτή είναι η ερώτηση. And last... Και ένα τελευταίο Θα είμαι γενή και θα σα ε, μεταφέρω άλλο ένα κουτσομπολιό. Κάτι που βέβαια είναι πολύ σημαντικό στο κοινοβούλιο, το κουτσομπολιό δηλαδή. Άκουσα ότι η διάσκεψη των Προέδρων το αξιοσέβαστο αυτό θεσμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο αποφάσισε φέτο να μην γίνει συζήτηση στην Ολομέλη για το προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Αυτό αποτελεί νεοτερισμό για το κοινοβουλευτικό έργο. Νομίζω ότι οποιαδήποτε έκθεση αξίζει να συζητηθεί στο, στο του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε την ποιότητα των συζητήσεων, αλλά ξέρετε, στον προβλησμό για να πω ιδίω στον προβλησμό, συνήθω οι συζητήσει που γίνονται είναι πολύ καλέ. Δίνουμε πάλι πυρομαχικά στου ε, λαϊκιστέ. Αν θέλουμε να εγκρίνουμε μια έκθεση χωρί συζήτηση, τι είδου κοινοβουλίου είμαστε τελικά αν ο ιστορικός κανονισμός προβλέπει συζήτηση πρώτης έγκρισης έκθεσης, θα πρέπει η συζήτηση να γίνει. Και έτσι είναι και το σωστό και για τον εισηγητή και για όλους όσοι στην Ολομέλη θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Πώς η διάσκεψη των Προέδρων και θα ήθελα να ξέρω και συγκεκριμένα ποια πολιτική ομάδα κατέθεσε αυτή την ε, ρηξικέλευτη πρόταση για να δούμε ποιοι είναι οι λαϊκιστές. Προσβλέπω λοιπόν κύριε Σιγητά μια καλή συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σβάλη, και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για τη σημαντική του δουλειά. Οφείλω να πω ότι ιδιαίτερα με ικανοποίησαν κάποια σημεία και θέλω να τα τονίσω στην ε, έκθεσή του. Συνεχίζω σε αυτό που στα Ταράντ σε σχέση με την δυνατότητα εξαγωγής συζήτησης στην Ολομέλεια, που για μας έχει θεμελιώδη σημασία η διεξαγωγή μιας συζήτησης με όλες τις πρακτικές δυσκολίες. Είναι απαραίτητο να γίνει μια συζήτηση για να προβληθούν ορισμένα βασικά προβλήματα που εντοπίζουμε σχέση με τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την αύξηση κατά 0,95%. Έχουμε μία πρόταση ακόμα χαμηλότερη εμείς και από την άλλη ο κύριος Δεπρέ μας λέει ότι υπάρχει δέσμευση για αύξηση του προϋπολογισμού που πρέπει να τηρηθεί σε σχέση με τους μισθούς βουλευτών και αποζημιώσεις βουλευτών και προσωπικού. Εμείς από την άλλη θεωρούμε ότι πρέπει αυτή η αναπροσαρμογή στον πληθω... με βάση τον πληθωρισμό να αναθεωρηθεί, γίνεται με βάση 11 χώρες και δεν λαμβάνει υπόψη το συνολικό πληθωρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον λαμβάνονται υπόψη χώρες που έχουν πολύ πιο υψηλούς ε, παράγοντες πληθωρισμού. Και άρα είναι δυσαναλογικά υψηλέ οι αυξήσει σε σχέση με την κατάσταση που ισχύει σε κάποια κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να ξανακοιτάξουμε αυτόν τον ε, κανονισμό και να θεωρήσουμε την κατάσταση αυτή. Επίση, ε, εγώ θεωρούσα ότι για, τις υψηλότερες, για τα υψηλότερα επίπεδα αποζημιώσεων αυτών των βουλευτών δηλαδή, θα ήταν καλό να σταματήσει, για τις αποζημιώσεις συγκεκριμένα των βουλευτών, να σταματήσει την αριθμική αναπροσαρμογή σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης. Είχε άλλωστε προταθεί, αν δεν απατώ, με να σταματήσει η αναπροσαρμογή για μισθού που ξεπερνούσαν ένα συγκεκριμένο ποσό του, 3.000 ευρώ ή κάτι τέτοιο. Πώ λοιπόν ζητούμε θυσίε από του πολίτε, όταν ιδιαίτερα για τόσο υψηλέ αποζημιώσεις και μισθούς ε, δεν προβαίνουμε σε, αντίστοιχα μέτρα. Ή θα ήταν αυτό καθήκον μα νομίζω για να δώσουμε και το καλό παράδειγμα ή εν πάση περιπτώσει πολιτικά να σταματήσουμε να απαιτούμε από τους άλλους να κάνουν οικονομίες όταν εμείς έχουμε ε, τόσο υψηλές αποδοχές και όταν ε, οι συντάξεις των απλών πολιτών που ξεπερνούν τις 3.000 δεν ακολουθούν την αναπροσαρμογή γιατί πρέπει οι δικές μας υποζημιώσεις που είναι ακόμη πιο υψηλές να την ακολουθούν. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από σταθμίσεις, γραμμικές σταθμίσεις, ε, περικοπές, συγγνώμη, σταθμίσεις περικοπές ε, στον προπολογισμό όπως κάθε χρόνο. Εδώ έχουμε να κάνουμε ζητήματα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης, που έχουν να κάνουν και με τις αποζημίωσεις των βουλευτών και τα γενικότερα ε, έξοδα που μπορούν να σχετίζονται με δαπάνες, των δαπανών των βουλευτών και εδώ μπορεί να γίνει μια περικοπή για να μειωθούν οι σχετικές δαπάνες. Για τις αποζημιώσεις όμως ταξιδιών θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιες λογικές ε, λύσεις, όπως σε τη οι διεισεξόδεις, να πραγματοποιούμε κάποια ταξίδια ή να εξασφαλίσουμε κάποιες συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες για πιο φτηνά εισιτήρια ή τη χρήση της οικονομικής ε, κατηγορίας, όπως πάντοτε εμείς υποστηρίζουμε, για τις μετακινήσεις μας. Και δεδομένου ότι έχουμε και την ε, κάρτα την ειδική. Μπορούμε ίσως να χρησιμοποιούμε το τρένο που θα μας έρχεται το ή άλλως δωρεάν. Γι' αυτό καλό θα είναι να, να προτιμούμε πάντοτε τις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές. Ιδίω για το, η μετάβαση στο αεροδρόμιο από εδώ εφόσον, ε, και εφόσον δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τις ειδικέ υπηρεσίες μεταφοράς του Κοινοβουλίου. Επίσης, καλό είναι να μην ε, χρησιμοποιούμε, όταν έχουμε τις δυνατότητες να χρησιμοποιούμε τα δικά μας μέσα για τις μετακινήσεις μας, δημόσιους πόρους για τις δαπάνες επικοινωνιακής πολιτικής ενώπιση των ευρωεκλογών. Είναι δυσανάλογα υψηλό το ποσό το οποίο προβλέπεται. Δεν αντιλαμβανόμεθα για ε, πώς θα αξιοποιηθούν ε, τα 25 περίπου εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται εδώ για την επικοινωνιακή πολιτική του Κοινοβουλίου. Θα θέλαμε μια ουδέτερη πολιτική, δηλαδή να μην υπάρχει προσπάθεια να προβάλλονται ορισμένες θέσεις και δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά όλες οι θέσεις και όλες οι ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια επικοινωνιακή πολιτική για το πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διαδικασία της συναπόφασης, ένα είδος πολιτικής αγωγής για τον πολίτη, ναι εντάξει μπορεί να υπάρχει ώστε να γνωρίζει καλύτερα το κοινό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά χωρίς να δίνουμε κατευθύνσεις πολιτικών επιλογών ή χωρίς να ε, εξέρουμε ορισμένες πολιτικές επιλογές που μπορεί ορισμένες πολιτικές δυνάμει ή ομάδες να μην θεωρούν σωστέ. Επίσης, ε, οι προβλέψεις για το ΚΑΔ, 14 εκατομμύρια για ένα τέτοιο έργο μου φαίνονται υπερβολικές, μας φαίνονται υπερβολικές και πρέπει να γίνει η περικοπή στις δαπάνες αυτές. Εν γέννη λοιπόν, ε, για να καταλήξω, θα κάνουμε τις σχετικές τροπολογίες για μας δεν πρέπει οι δαπάνες να ξεπερνούν δεν πρέπει να ξεπερνούν τις περσινές, δεν πρέπει να υπάρξει αύξηση. Αντιθέτως, μείωση θέλουμε να δούμε και πάντως θέλουμε από το 2019 μια αναθεώρηση ορισμένων βασικών αρχών και κυρίως την αναποσαρμογή με στον τιμάριθμο και γενικότερα περικοπές ε, ίσως με κάποια σταδιακή ε, μείωση από το 2019. Από το 2009 ήδη έγιναν κάποιες αλλαγές. Δέκα χρόνια μετά νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο προς την ίδια κατεύθυνση για περικοπή των δαπανών και αναθεώρηση ορισμένων ζητημάτων και ε, λύσεων έτσι ώστε να δώσουμε και στον πολίτη πιστικά την εικόνα ότι προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία όσο δυνατόν από την δαπάνη δημοσίων πόρων. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Σάνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, καθώς οι συνάδελφοι σήμερα αρκετά θέματα ήδη. Ενώ όλο το κείμενο που είδαμε συνιστά μια καλή βάση εκκίνησης και τη γοφρονώ ότι υπάρχει ακόμη δουλειά για ορισμένα σημεία Εν γέννη σημειώνω πως δεν συμφωνώ με τα όσα είπαν κάποιοι συνάδελφοι. Ο προπολογισμό ε, εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι όλα οι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζονται σαν να είναι τέλειες. Ε, δεν συμφωνώ λοιπόν. Αντιθέτως βλέπω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για βελτίωση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουμε, όπως μπορεί κάποιος να πιστέψει, να, ε, καταστρέψουμε τις, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αντιθέτως θέλουμε να λειτουργήσουν καλύτερα, να βοηθήσουμε να λειτουργήσουν καλύτερα και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, μια προσέγγιση θετική και ενώπιον του πολίτη. Εάν μπορούμε να δαπανούμε καλύτερα τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου και εκείνος θα είναι πιο ικανοποιημένος και εκείνος θα θεωρήσει ότι τα θεσμικά όργανα λειτουργούν καλύτερα. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό να έχουμε, και θα έχουμε θετική ανταπόκριση πιστεύω. Ε, τα σημεία στα οποία χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Και θα σημειώσω ότι δεν θεωρώ ότι η έλλειψη συμμετοχής ή η απώλεια η απουσία γνώσης ή η απόσταση που έχει ο πολίτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν απόρρια ε, περιορισμένων δαπανών ή περικοπών ή λιγότερων επενδύσεων. Αντιθέτως, νομίζω, οφείλονται σε μια εσφαλμένη διαχείριση σε νόμους ε, που εγκρίναμε εμείς εδώ και που δεν ενέκρινε ο πολίτης. Θεμελιώδες, λοιπόν. Πρώτον, για την επικοινωνιακή πολιτική και τις σχετικές δαπάνες χρειάζεται να έχουμε στο δυνατόν πιο ευρεία κάλυψη και ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή όπου τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία και ο πολίτης έχει όλο και μεγαλύτερη απόσταση και δυσπιστεί απέναντί τους δαπάνες επικοινωνιακής πολιτικής από τα θεσμικά όργανα και προτάσεις όπως αυτές που είδαμε για τις ευρωεκλογές του 2019 από πλευράς της γραμματείας μοιάζουν περισσότερο σαν μια απόπειρα τα κονδύλια αυτά να τα χρησιμοποιήσει κανείς για προπαγανδιστικούς σκοπούς σαν να προσπαθεί να κρατηθεί από ένα σωσίβιο πριν πνιγεί, το σωσίβιο της ε, επικοινωνιακής πολιτικής. Ε, δεν ε, θα τα καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο, να, τρόπο να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή του πολίτη στις ευρωεκλογές. Μόνο αν έχουμε καλό νομοθετικό έργο με νομοθετικά κείμενα αποτελεσματικά κατανοητά. Και αυτό άλλωστε έχουμε προτείνει και με τις τροπολογίες μας που είναι απολύτως αντίθετες στην προσέγγιση ε, που προβάλλεται σε σχέση με τις επικοινωνιακές δαπάνες για τις εκλογές του 2019. Σε σχέση με άλλες ε, προτάσεις, άλλα σημεία, θεωρώ πως πρέπει να κοιτάξουμε με πολύ πιο προσεκτικό τρόπο την πολιτική τη σχετική με τα κτίρια και εδώ γίνονται ε, διάφορες αναδιαρθρώσεις, ε, φτιάχνονται καινούρια κτίρια από το μηδέν ή καταστρέφονται παλαιά κτίρια για να ανοικοδομηθούν ε, θεμελίων. αλλά νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε πολύ περισσότερη λογική όλη αυτή την ιστορία της κτηριακής πολιτικής, γιατί η μέση, η διάρκεια ζωής ενός ε, κτηρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαίνεται να μην ξεπερνάται 25 χρόνια. Λίγο μάλλον μου φαίνεται. ας το κοιτάξουμε λοιπόν και αυτό κατά τρόπο ορθολογικό και ας προσπαθήσουμε με την συντήρηση να ε, παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής των κτηρίων μας. Και όπως ε, επεσήμαναν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι νωρίτερα, ας βεβαιωθούμε ότι με την χρήση νέων τεχνολογιών και νέων μέσων επικοινωνιακής πολιτικής θα μπορούσαμε να μειώσουμε ακόμη και τους χώρους που χρειαζόμαστε. Και άρα και τα κτίρια. στα μέσα για την ασφάλεια. Πολύ σημαντικά ασφαλώς στην εποχή που ζούμε. Ο, Ευρω... ο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ενισχυθεί σημαντικά στον τομέα αυτό. Αλλά και εδώ βλέπω ότι κάποιες δαπάνες μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή δυσνόητες. Πρόσθετο προσωπικό για την ασφάλεια, Φερρυπίν. Ένοπλο προσωπικό για την ασφάλεια και επιπλέον προσωπικό για την ασφάλεια του ίδιου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δίνεται η εντύπωση ότι μάλλον θέλουμε να κλειστούμε παρά να ανοίξουμε προς τα έξω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά υπάρχει ένα κονδύλιο που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα να επανεξετάσουμε τις δαπάνες συγκεκριμένα των πολιτικών ομάδων, γιατί κάθε χρόνο διαπιστώνεται ενίσχυση των δαπανών, των πόρων που διατίθενται στις πολιτικές ομάδες, είτε για το προσωπικό τους, είτε για τη λυπή χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση σε κόμματα και ιδρύματα ευρωπαϊκά έχουν αυξηθεί κατά 250% από το 2008 μέχρι σήμερα. Πρόκειται για τις δύο γραμμές του προϋπολογισμού που παρουσιάζουν την υψηλότερη αύξηση στην περίοδο αυτή. και νομίζω ότι τα ποσοστά αυτά ξεπερνούν κατά πολύ τον προπολογισμό, τον ε, πληθωρισμό, συγγνώμη. Άρα πρέπει να περιορίσουμε τι δαπάνε αυτέ. Βεβαίω, είναι σαφέ ότι στη δημοκρατία πρέπει όλοι να τη χάνουν τη ίδια χρηματοδότηση, ισότιμη χρηματοδότηση, για να έχουν τη δυνατότητα να ακουστεί και η φωνή του σε πολιτική. Αλλά πρέπει να συγκρατήσουμε και να εξισορροπήσουμε κάπω τα νούμερα αυτά. Πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε πάνω απ' όλα. Το ίδιο και για το προσωπικό που ανέφερε και ο κύριος Ταράντ. Επιπλέον 76 θέσεις προσωπικού για τις πολιτικές ομάδες μέσα στην τελευταία χρονιά. Και έχω ζητήσει εγώ συγκεκριμένε διευκρινήσεις για τους 50 AST θέσεις βοηθών, βοηθητικού προσωπικού που μετατρέπονται σε ε, προσωπικό διοικητικό, AD. Γιατί και πώς και τι κόστος θα έχει όλο αυτό. Mm. Κόστος οικονομικό και λειτουργικό. Τελευταία παρατήρηση. Σχετική με το πώς θα μπορούσαμε να εξορθολογήσουμε άλλες δαπάνες. Ο κύριος Δεπρέ είπε όντως ότι ε, κάποιες από τις δαπάνες ε, που αναφέρονται στο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν να κάνουν με αυξήσεις που ακολουθούν τον αντιμάριλθμο. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία και να μην προσπαθούμε να βρούμε στον κατάλληλο τόπο τις λύσεις για εκείνες τις δαπάνες οι οποίες δεν μας επιτρέπουν μια ευελιξία στη διαχείριση του προϋπολογισμού αν πάνω από το 60% των δαπανών είναι αναπροσαρμοσμένες στον τιμάριθμο δεν μπορούμε να τις πειράξουμε και άρα η δουλειά μας είναι ακόμη πιο δύσκολη. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να καταστήσουμε πιο ευέλικτες τις λοιπές δαπάνες έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και περικοπές λιγότερο γραμμικές, πιο ουσιαστικές χωρίς να πληγούν κάποιες γραμμές του προϋπολογισμού που θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν σε κάποιες παραμέτρους. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την διαχείριση της ε, έκθεσης από τον εισηγητή. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλή συνεργασία. Ελπίζουμε και με τη γραμματεία. Και ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Ευχαριστώ. Thank you very much. I see no other colleagues wanting... Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο άλλο συνάδελφο το λόγο. Να δώσω στον κύριο Κλέφη τη δυνατότητα να πάρει το λόγο γάμα δέλτα από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Νίκο Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Απόψε λαμβάνει η χώρα η πρώτη συνδιαλλαγή μεταξύ μελών του Προεδρείου Γενικής Γραμματείας ε, ημών και των ε, προπολογισμών. Νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα όπως αυτά που είπε ο κύριος Ντεπρέ για την χρηματοδότηση του κτηρίου ΚΑΝΤ στο Λουξεμβούργο, Κόντραντ Αντενάουρ. Υπάρχουν ε, κάποιες διευκρινήσεις που πρέπει να δώσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Το δημοσιονομικό κονδύλιο που πρικοδοτείται στην αρχή του έτους ε, στόχο έχει να χρηματοδοτήσει την προετοιμασία των έργων, ουσιαστικά δηλαδή μελέτες και φύλαξη του εργοταξίου. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτό το οποίο χρησιμοποιούσαμε για το ράμα το λεγόμενο ήταν ε, τα έργα, αυτά καθεαυτά. Θα έχετε έτσι λοιπόν μια ξεκαθαρή εικόνα για το τι απομένει να χρηματοδοτηθεί για το Conrad Adenauer, ποιε είναι οι εναλλακτικέ και θα λάβετε πιστεύω τη δέουσα πολιτική απόφαση έχοντας υπόψη και τα στοιχεία και τα πολιτικές παραμέτρους. Ε, κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά το ποσοστό δημαρχημικής αναπροσαρμογής, το συντελεστή, χρήσιμο πιστεύω είναι να τηρούνται οι κανόνες που ισχύουν. Βέβαια γνωρίζουμε ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί μπορούν να εξελιχθούν και να τροποποιηθούν σε ό,τι αφορά τις αποδοχές των βουλευτών, ε, των συνεργατών, του προσωπικού, των ε, συμβασιούχων. Οι απολαβές αυτές ε, έχουν οριστεί βάση μεθόδου, την οποία προβλέπει το καταστατικό. Και γίνεται ένας στατιστικός υπολογισμός που εσείς ίδιοι ως νομοθέτες έχετε καθορίσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ισχύει ο κανόνας. Μέχρι όταν να ο εν λόγω κανόνας, και επαναλαμβάνω εσείς είστε αρμόδιοι, οι συνομοθέτες, εσείς και το Συμβούλιο, αφού πρόκειται για διαδικασία στην απόφαση, στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει τον κανόνα αυτόν τον σεβαστούμε. Υπάρχει υποχρέωση να τηρήσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά το γενικό δίκτυο πληθωρισμού. Δεν χρησιμοποιούμε το ε, δίκτυο πληθωρισμού εξάντε για την κατάρτιση του προβλησμού. Βλέπουμε κονδύλι ανακονδύλιο το δίκτυο που θα εφαρμόσουμε. Επενθύμησε ο κύριος Δεπρέ ότι σχεδόν για το 60% έχουμε αυτή την περίφημη γνωστή μέθοδο σε σχέση με τη μισθολογική εξέλιξη για το προσωπικό, για βουλευτές και συνεργάτες, για άλλα κονδύλια. Μετράει ο τόπος εργασίας κυρίως. Αν τα κτίρια βρίσκονται σε Στρασβούργο, Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή στη συγκεκριμένη ε, πόλη λαμβάνεται υπόψη και όχι τι ισχύει σε μια άλλη χώρα πιο μακριά. Αναλύουμε λοιπόν κάθε κονδύλιο ξεχωριστά για να δούμε κατά πόσον προκύπτει ε, τη μαριθμική αναπροσαρμογή, ανάγκη τη μαριθμικής προσαρμογή Δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Συλλογικά όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη για την κατάρτιση του επόμενου προπολογισμού. Και αν συγκρίνεται αυτό το προηγούμενο με το προηγούμενο, διαπιστώνεται ότι υπάρχει αύξηση. Διαπιστώντα ότι υπάρχει αυτή η αύξηση, κινούμε έχοντας ως ένα στοιχείο πιθανής ανάλυσης το δίκτυο πληθωρισμού. Ε, δεν είναι εξάντε, επαναλαμβάνω όμως αυτός ο υπολογισμό απλά διαπίστωση των περιορισμών. Στο ό,τι 25 εκατομμύρια που προβλέπονται για την προεκλογική εκστρατεία της ευρωεκλογής, ε, φυσικά πρόκειται για έκτακτη δαπάνη, υπό την έννοια ότι επί τετραετία αυτή δαπάνη δεν υπάρχει αν το κοινοβούλιο θέλει κάποια στιγμή να κινητοποιήσει διάφορα εργαλεία, ο κ. Ντεπχέ σωστά είπε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα πλέον σύγχρονα εργαλεία. Θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση σε βάθος ε, για τη στόχευση και για το ποιοι είναι αυτοί που δεν είχαν τόσο πολύ ε, ενημέρωση από το Κοινοβούλιο. οι πολίτες πρέπει να έχουν αντίληψη ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψήφο τους ε, για να καθορίσουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξασφαλίσετε εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να ενημερωθούν οι πολίτες. Για τις πιο πολιτικές αποφάσεις νομίζω ότι καλό είναι να περιμένετε την ε, συζήτηση που θα έχετε στη συνέχεια με τα μέλη του Προεδρείου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάφη και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ήταν πολύ επικοδομητικά και πολύ πλούσια η συζήτησή μας. Ένα-δυο σχόλια δικά μου πριν που κλείσουμε προς τον Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες να το επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι θα πανούμε μόλις 6% του προπολογισμού για διοικητικές δαπάνες. Δίκιο έχει, έτσι είναι, σε κάθε τομέα της ζωής. Δημόσιο, ιδιωτικό, όταν έχουμε να κάνουμε με πελάτες, καταναλωτές, κοινό. Η κάθε οργάνωση οργανισμός πρέπει να κοιτάζει προσεκτικά εάν περνάει όχι το όριο του 6%. Δέχομαι το σχόλιο σας, διότι όντως δεν υπάρχουν πολλοί δημόσιες φορείς, πολλοί δημόσιοι φορείς που να ε, ακολουθούν το παράδειγμα του Κοινοβουλίου. Βεβαίω, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει υποστηθέμενη αξία. Δηλαδή τα χρήματα που δαπανούμε ότι κάτι προσφέρουν. Σωστά επενθυμίστε και ότι πάνω από τα δύο τρίτα των δαπανών του προπολογισμού είναι ήδη σταθερέ. Και υπολογίζονται με συντελεστή. 30% του προπολογισμού ε, κατευθύνεται προ τι αποταμιεύσει. Κάποιοι ενδιαφέρον επίση στην ε, διαφάνεια, με την οποία συμφωνώ απολύτως. Και πολλοί μίλησαν για κόμματα και ιδρύματα. Και κάποιοι το ανέφεραν και στο επίπεδο των γενικών δαπανών. Ως ε, εισηγητής θα δείξω διαλεκτικότητα για το επίπεδο των δαπανών. Απλώ και τα σχόλια του κυρίου Τζάνι τα λαμβάνω υπόψη για την αύξηση από το 2008 52 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σήμανε. Το συνειδητοποιώ αυτό, αλλά ταυτόχρονα τα γεγονότα των τελευταίων δύο ετών και τη τελευταία ειδικά χρονιά δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιε αδυναμίε στον έλεγχο των ταπανών, ε, της, δημοκρατικού ελέγχου δηλαδή για το πώ ταπανήθηκαν τα χρήματα αυτά. Θα πρέπει να ισχύσουν διαδικασίε ώστε την επόμενη θητεία να έχουμε πιο ε, ασφαλείς διαδικασίε για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει. Ευχαριστίες προς τον κύριο Ντιπρέη που μου θυμίζει και πάλι τη σημασία των αριθμών. Το 1,7% ως προς το πληθωρισμού που δεν θέλουμε να το υπερβούμε, σωστά το άκουσε και το είπα, αλλά θα ξέρετε στην αρχική πρόταση οι αριθμοί με τους οποίους ξεκινήσαμε ήταν το 0,95%. Ξέρω όμω, Ζεράρο, ότι θα έχει ενεργικό ρόλο στις δημοτεύσεις που θα ακολουθήσουν ούτως ή άλλως. Επίσης για το Ρεμασάζ θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τους τίτλους όπου υπάρχει λιγότερη δαπάνη από αυτή που αρχικά προβλεπόταν και τα ποσά που περισσεύουν. Για τη στρατηγική των κτηρίων, πολλοί συνάδελφοι σχολίασαν αυτό το θέμα. Σημειώνω τα όσα είπαν και περιμένω περισσότερες πληροφορίες από το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα διευκρινίσει περισσότερο, ελπίζω, καθώς θα προχωρεί η εκπόνηση της έκθεσης, πώς δαπανώνονται τα χρήματα και πού ακριβώ. Για τι ερωτήσει του κυρίου Τάραντ. Το θέμα των βοηθών, των τοπικών βοηθών, των διαπιστευμένων βοηθών Θα συμφωνήσω ότι υπάρχει ανάγκη διευκρίνηση, τα είπε και ο κύριος Ντουσάντου, αλλά είναι σαφές, εδώ δεν επιζητούσε να διευθετήσω τις πληρωμές προς τους βοηθούς, απλώς κάποια αποσαφήνιση χρειάζεται, διότι υπήρξαν περιπτώσει, όπου η έλεγχη ήταν κάπως αδύναμη. Ο αριθμό των βοηθών που απασχολώνται στην ε, χώρα προέλευση αυτού που, ονομάζουμε ε, τοπικούς, φαίνεται υπερβολικό. Χρειαζόταν κάποια αιτιολόγηση σε κάποιε περιπτώσει. Εκεί λοιπόν επέστησα την προσοχή τη Επιτροπή στο γεγονό ότι χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση. Και επίση ιδιαίτερα με ε, αφορούν τα θέματα για τα επιδόματα και τα περντίεμ του Στρασβούργου. Ναι, θα φροντίσω και αυτέ οι ανησυχίε να βρουν τη θέση του στην έκθεση. Και προ τον κύριο Τάραντ και τον κύριο Βάλλη, δίκιο έχετε. Τα συζητήσαμε και στην Ολομέλεια και πιστεύω ότι η βασική αρχή των ε, δημόσιων ε, λογαριασμών είναι ακριβώ η διαφάνεια. Αυτή η πρέπει που διαπνέει. Και είναι περίεργο που δεν θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια. Ε, η συνδιαλλαγή, που σα είπα, είναι προγραμματισμένη σήμερα. Το γνωρίζετε. Είναι στι 6.30. Στι 3 Απριλίου θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών στο Στρασβουργό και στις 5 ή 6 Απριλίου η έκθεση θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Σε αυτή τη φάση να πω ότι έφτασε ο Πρόεδρός μας, χαίρομαι πολύ γι' αυτό, τον προσκαλώ να λάβει τη θέση του στο Προεδρείο και κλείνω τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν παρόν στις τρεις ε, οπότε και ξεκίνησε η συνεδρίαση, μια άκρο σημαντική συνεδρίαση. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Άσχουρθ ε, που χρημάτισε πρόεδρος, αλλά ήταν και συγητής για το σχέδιο προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι προοδεύουμε σε θέματα διαφάνειας ε, παρουσίασης του προβλέψιμου του Κοινοβουλίου, αλλά υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Αφού σας ευχαρίστησα και είπα και όλα αυτά, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Έτιγκερ που με την παρουσία του μαρτυρά πόσο δεσμευμένο είναι στο να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή Προπολογισμού. Σα ευχαριστώ πολύ, ειλικρινά, για την παρουσία σα εδώ, κύριε Επίτροπε. Θα μιλήσουμε εκ νέου για το σχέδιο ενδιάμεση αξιολόγηση του πολιτου δημοσιονομικου δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Είναι σημαντικό, είναι σημαντική αυτή η χρονική στιγμή, ε, επί εβδομάδε Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση από το Συμβούλιο. Τώρα φαίνεται ότι η Ιταλική επιφύλαξη ήρθε. Επομένως, θα πρέπει να αποφασίσουμε για το κατά πόσον είναι σκόπιμο ή όχι να δώσουμε την σύμφωνη γνώμη μας για αυτό το σχέδιο αναθεώρησης, επανεξέτασης. Να δώσω το λόγο αν συμφωνείτε πρώτα απ' όλα στους συνεισηγητές. Η κυρία Τωμά καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο συνεισηγητής μου ε, έχει πρόβλημα διότι καθυστερεί πτήση του. Ο κύριος Φερνάντες ίσως θα πάρει το λόγο ανταυτού. Θα προσπαθήσω εγώ να κάνω μια σύνοψη της κατάστασης. Ε, εν συντομία λοιπόν να σας πω, τον Ιούλιο του 2016 αν θυμάστε, υιοθετήσαμε στο Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, με φιλόδοξη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Η δυνατότητα αυτή μας ε, δίνεται στο πλαίσιο αυτό ε, της περίοδου 2014-2020. Η εξέταση λοιπόν του προϋπολογισμού και του πολίτου πλαισίου αναλυτικά. Έπειτα είχαμε το σχέδιο θεώρηση από την Κομισιόν και τον Νοέμβριο ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις παράλληλα με το προπολογισμό. Θεωρούσαμε ότι πράγματι θα μπορούσαμε να προβούμε στην απαιτούμενη αξιολόγηση, αναθεώρηση μάλλον. Δεν ήταν απλές οι διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Έγινε παρόλα αυτά μια πρόταση που ήταν και παραμένει χαμηλότερη κατ' εμέ των αναγκών και εμείς ε, επιχειρηματολογήσαμε υπέρ της ανάγκης ε, αναθεώρησης. Και στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό ήμασταν κοντά στην επίτευξη αποτελεσμάτων, παρότι δεν συνέπεπταν οι απόψεις μας με αυτές του Συμβουλίου. Υπήρχε και η Ιταλική επιφύλαξη που προσέγγιζε τις δικές μας επιφυλάξεις. Πριν από 15 μέρες ήρθε αυτή η Ιταλική επιφύλαξη. Προτείνει τώρα λοιπόν αναθεώρηση το Συμβούλιο με αύξηση το μηχανισμό ευελιξίας, αφενός τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τα αδαπάντα κονδύλια του Ταμείου Προσαμής στην Παγκοσμιοποίηση και του Ταμείου αλληλεγγύης Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο αυτή τη ευελιξία. Επίση, προτείνει την μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τα κονδύλια μετανάστευση ασφάλεια και μία αύξηση του ανώτατου ορίου για τις πιστώσεις πληρωμών, τρία δι συνολικά όλα αυτά. Η πρόταση αναθεώρησης συνδέεται με τέσσερις ε, δηλώσεις του Συμβουλίου, τις οποίες μας προτείνει το Συμβούλιο να επικυρώσουμε από κοινού. Έχουμε μια δήλωση που δεν μας δημιουργεί πρόβλημα, Τεχνική φύσεως θα τη χαρακτήριζα. Έχουμε μία δήλωση για την παρακολούθηση του στόχου μείωση ε, του προσωπικού κατά 5% για το προσωπικό του κοινοβουλίου ή μάλλον συνολικά των θεσμικών οργάνων. Υπάρχει μια δήλωση και σε αυτήν θα επιμείνω λίγο. Περιλαμβάνει ενισχύσει και κάποια όρια και ε, επαναχρησιμοποίηση κάποιων κονδυλίων αναφέρεται πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ε, πέραν ε, των 500 εκατομμύρων προβλέπονται στο προπλησμό 2015. 700 εκατομμύρια, 1,4 δις, 1,2 ε, την ασφάλεια. Αυτά έχουν ας πούμε επικυρωθεί και μια ένδειξη ότι στο 1α για την ανάπτυξη την απασχόληση θα δοθούν κάποια εκ νέου κονδύλια. 2,8 δηλαδή δις ευρώ. Φρέσκο χρήμα, 6 δις, εκ των οποίων για τα τρία θα χρειαστεί απόφαση των δύο σκελών της Δημοσιονομικής Αρχής, της Αρχής επί του Προπολογισμού. Η τελευταία αυτή δήλωση συζητήθηκε πολύ γιατί θα μπορούσε να θεωρηθεί περιορισμός των αιτήσιων συζητήσεων ε, μεταξύ Συμβουλίου Κοινοβουλίου για το προϋπολογισμό. Θα μπορούσε, λέω. Δεν μπορούμε να επαξοφλήσουμε την ερήσια δημοσιονομική συζήτηση και τις ε, αρμοδιότητες ε, των σχόλων του προϋπολογισμού πέραν της αναθεώρησης και των δηλώσεων, εμείς προτείνουμε και μια άλλη δήλωση, η οποία εκπηγάζει από το Κοινοβούλιο αυτή τη φορά, η οποία λοιπόν ερμηνεύει και διευκρινίζει τις δηλώσεις του Συμβουλίου. Διότι φυσικά και ικανοποίηση μόνο μπορεί να προκαλέσει το γεγονός ότι Όταν ξεκινήσαμε ε, στην Επιτροπή Προπολογισμών ε, φαινόταν να μην υπάρχει προσέγγιση παρά ε, τα αντίθετα προγνωστικά φτάσαμε σε αυτή τη θέση του Συμβουλίου άρα δεν θα ήταν σκόπιμο να μην επικυρώσουμε πιστεύω αυτήν την αναθεώρηση που δεν φαινόταν καθόλου πιθανή αρχικά την επικυρώνουμε βέβαια δεχόμαστε και τις δηλώσεις αλλά όπως είπα θα θέλαμε να προσθέσουμε μία δήλωση του Κοινοβουλίου που θα διευκρινίζει την ερμηνεία των δηλώσεων και της τελευταίας που σας ε, εξέθεσα αναλυτικότερα. Θα μπορούσε να θεωρείται υποχρέωση για περιορισμό των νησίων τα top-up ε, ή για το redeployment. Θέλουμε λοιπόν με αυτή τη διευκρινιστική δήλωση να αναφέρουμε ότι αυτές οι κοινέ δηλώσεις δεν έχουν καμία ε, νομική υποχρέωση, δηλαδή το Κοινοβούλιο παραμένει ελεύθερο να αποφασίσει. Ορίστε. Να προσπαθήσει, λέει ο κ. Ντεπρέ. Παραμένετε αισιόδοξο, αθεράπευτε αισιόδοξο, κ. Ντεπρέ. Τέλο πάντων, ναι, να προσπαθήσει να αποφασίσει για την ετήσια εξέλιξη του προπολιτισμού Δεύτερον, να υπενθυμίσει το Κοινοβούλιο ότι θα ασκήσει τι προνομίε του ε, στο απόλυτο, εξάρτηση οποιασδήποτε δήλωση και επίση ε, για το redeployment αυτό θα αφορά μόνο προγράμματα κλειδιά, μόνο εφόσον ευνοούν όμω την ανάπτυξη, την απασχόληση για την κάλυψη των ε, πιεστικών αναγκών του σήμερα και εφόσον υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό εκτέλεσης. Σε αδρές γραμμές αυτές είναι οι προτάσεις που διατυπώνουμε ο Γιάνν Όλμπριχτ και εγώ σήμερα για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε, αν θέλετε, αυτή την πρώτη αναθεώρηση του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου. και να διατηρήσουμε ε, τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες ε, που έχει το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε κυρία Τωμά για αυτήν την ε, πρόταση για να γίνει αδιαμφισβήτητα κάποια πρόοδος και να μπορέσει το Κοινοβούλιο να βρει μια προσέγγιση σταθερή. και να καταπιεί το πικρό ποτήρι των statements. Έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν δυσκολίες για τον συνάδελφο ε, με τις ε, αεροπορικές μεταφορές. Θα δώσουμε την ευκαιρία στον κύριο Φερνάντες να τον ε, αντικαταστήσει. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του συναδέλφου και συνεισηγητή για την αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου θα ήθελα να λάβω το λόγο αλλά και για προσωπικούς σκοπούς για να υποστηρίξω τους δύο συνεισηγητές και να τους συγχαρώ για την εξαιρετική τους δουλειά για την ε, φιλοδοξία που έχουν θέσει στους στόχους και για το αποτέλεσμα που έχουν επιτύχει ως τώρα. Να ξεκινήσω θυμίζοντας και στον Επιτροπό μας, στον οποίο χαιρετώ, ότι το Κοινοβούλιο στις Δημοτεύσεις του Πολιτικού Δημοσιονομικού Πλαισίου ζήτησε τη δυνατότητα της ευελιξίας και τη δυνατότητα αναθεώρησης. Αγωνίστηκε για αυτό το σκοπό πολλές φορές παρά την βούληση του Συμβουλίου και για τα δύο αυτά σημεία. Και παρόλα αυτά τώρα καταφέραμε να υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης και ευελιξίας. Περάσαμε όμως από πολλά κύματα στην Ένωση, ιδίω με το θέμα των ε, προσφύγων. Θα ήταν καταστροφική η απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άποψη του προπολογισμού αν είχαμε μείνει στην αρχική πρόταση. Γιατί όμως πρέπει πάντα το Κοινοβούλιο να είναι το θεσμικό όργανο που πάντοτε απαιτεί περισσότερη ευελιξία, που πάντοτε απαιτεί καλύτερη διαχείριση των πόρων και είναι το πιο υπεύθυνο ως προς αυτά. Ενώ το Συμβούλιο θα έπρεπε να επιδιώκει τα ίδια συμφέροντα. με το 80% των ε, ε, πόρων μας. Αυτή η αναθεώρηση λοιπόν είναι η δυνατότητα να δώσουμε μια καλύτερη απόκριση στα προβλήματα των πολιτών, στα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις προκλήσεις που βιώνουμε. Και χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς καμία διάθεση να χρυσώσει το χάπι, θα έπρεπε να είναι αυτή η στάση και του Συμβουλίου. Αυτήν την ευελιξία που ζητούσαμε επιτυγχάνουμε τώρα. Θα είχαμε προβλήματα με τις πληρωμές. Θέλουμε να αποκριθούμε στους στόχους της ανάπτυξης και την απασχόληση, την απασχόληση ιδίως των νέων. Μπορούμε επιτέλους τώρα να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία χωρίς εμπόδια για το συνολικό περιθώριο των πληρωμών και το γεγονός ότι ε, ενισχύθηκε το εργαλείο της ευελιξίας και το περιθώριο για τις απρόβλεπτες ανάγκες ή το Ταμείο της Αλληλεγγύης και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και η δυνατότητα να ανατρέξουμε σε αυτά, όλα αυτά είναι θετικά σημεία. Θετικά σημεία τα οποία θα επιβεβαιωθούν στη μελλοντική εκτέλεση. Και είναι και θεμελιώδου σημασία όλα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την διαχείριση του υπολογισμού. Ελπίζω να μαλοχαιρετώ την ομοφωνία του Συμβουλίου και θα έλεγα κιόλα επιτέλου. Καιρό ήταν να φτάσει το Συμβούλιο σε αυτή την ομοφωνία. Ήταν καιρό να το πετύχουμε κι αυτό. Όμω το Συμβούλιο ανέκαθεν είχε και ακόμη έχει τον πειρασμό να προσπαθήσει να δέσει τα χέρια του Κοινοβουλίου όσο μπορεί. Και αυτός ο στόχος πολλές φορές είναι ακατανόητος. Το Κοινοβούλιο είναι ένα θεσμικό όργανο που είναι σύμμαχος του Συμβουλίου. Και τώρα φτάνουν αυτές οι δηλώσεις. Οι δηλώσεις που δεν έχουν αξία νομική. Δεν είναι δηλώσεις θα έλεγα, που δεν αφήνουν ευελιξία, την κάνουν ακόμη πιο δεδομένη. Οι πολιτικές δηλώσεις δεν υπερισχύουν των συνθήκων. Οι πολιτικές δηλώσεις δεν υπερτερούν των διαδικασιών του προπολογισμού. Είναι προφανές. Στα θέματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέταση, όπως η αναθεώρηση, μάλλον καλυτερη παράταση της χρήσης ε, και της εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Θετικές επενδύσεις, του γνωστού προγράμματος Juncker και όλων των άλλων νομοθετικών θεμάτων που αυτή τη στιγμή εξετάζονται τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει ότι λόγω των δηλώσεων αυτών εμεί θα χάσουμε τα προνομιά μα και τι αρμοδιότητέ μα. σα ίσα στην ίδια την κοινή δήλωση βρίσκεται η απάντηση. Αυτό που είναι κατάφορο και προφανέ, πρόδειλο μάλλον και προφανέ, είναι ότι οι ίδιε οι δηλώσει δεν θέτουν ένα αμφιβόλο τις αρμοδιότητες και τα προνόμια της δημοσιονομικής αρχής. Έτσι, Υπογράφουμε και εμεί αυτέ τι δηλώσει και κάνουμε και εμεί από την πλευρά μα μια άλλη δήλωση, όπω είπε και η κυρία Τωμά, για να διευκρινίσουμε του όρου τη δική μα ε, τοποθέτηση. Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι ότι αυτή η επιτυχία, αυτή η δυνατότητα που προηγουμένω δεν προβλεπόταν και δεν ε, προστατευόταν στο πλαίσιο του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, αυτή η πρώτη αναθεώρηση του Πουδουπού είναι ένα μήνυμα μπορούμε να έχουμε ένα καλό πλαίσιο και μετά το 2020. Αυτό ανέκαθεν ήταν ο στόχος του Κοινοβουλίου. Να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ευελιξίας. Και με κάτι άλλο κατά νου. Να μην χάσουμε ε, και τις, ε, τα, τα κονδύλια, ούτε ένα λεπτό του ευρώ, από τις ε, δεσμεύσεις για πληρωμές του προϋπολογισμούς του προπολογισμού. Θέλουμε να επιδιώξουμε τους στόχους της Στατικής Ευρώπη 2020, να κοιτάξουμε τα προβλήματα που μας δημιουργούν η μετανάστευση, οι πρόσφυγες, η τρομοκρατία, η ανάγκη για να τονωθεί η ασφάλεια, να έχουμε καλύτερη άμυνα και κοινή άμυνα. Η παρουσία του Επιτρόπου εδώ είναι μια εγγύηση. Εγγύηση ότι θα εργαστούμε από κοινού για να πετύχει όχι μόνο η αναθεώρηση αυτή στην υλοποίησή της, αλλά και για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για να είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Merci, monsieur le rapporteur général. Ευχαριστώ τον Γενικό εισηγητή για το 2016 που μετέφερε και τα λόγια του κυρίου Ολμπριχτ. Και θα ακούσουμε τώρα την Επιτροπή με τον κύριο Έτσιγκερ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Η ενδιάμεση αναθεώρηση έχει ιστορικό χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο συμφωνείται από την αρχή της διαρκείας μεταξύ Συμφωνίου, Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής να γίνει αναθεώρηση στο μισό της διαδρομής και να υλοποιηθεί αυτή. Και πρέπει να επενέσουμε ρητά το Κοινοβούλιο. Ήταν δική σας η ιδέα αυτή. Στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δηλαδή να διατηρήσετε την επιρροή. Κάνατε την διαπραγμάτευση το 2013 σκληρά, προχωρείτε και αυτό το αφήνουμε όλα σε εσά. Η κυρία Τόμας και ο κύριος Όλμπριχτ, οι δύο συνεισηγητές με την εκπροσώπηση του κυρίου Φερνάντες συγκεκριμένα έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και πολύ καλή ήταν και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε επίπεδο. Στο Συμβούλιο από τα μέσα Νοεμβρίου ως αρχάς Μαρτίου έγιναν διαβουλεύσεις. Διήρκεσαν αρκετά δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι ήταν αρκετά μακρά η διαβούλευση επί Συμβουλίου, ε, το Κοινοβούλιο και διατήρησε την, ε, ε, τις θέσεις του, αλλά και δούλεψε γρήγορα και με αποτελεσματικότητα και πολύ καλή γνώση του θέματος και χρησιμοποιεί αυτό το χρονικό παράθυρο ώστε να ενσωματώσει και ζητήματα που προκύπτουν από την επίκληση του άρθρου 50 από το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτό το ενδιάμεσο διάστημα και να τα εγγράψει σε όλα τα θέματα του προϋπολογισμού. Είναι ανοιχτό λοιπόν αυτό το παράθυρο, το χρονικό παράθυρο, χωρί όμω να μπορεί κανεί να πει ότι θα κρατήσει και για πολύ μεγάλο διάστημα. Γι' αυτό θα, είναι πολύ, ήμουν πολύ ευγνώμων ε, προ τον Πρόεδρο και του συζητητέ αλλά και τι πολιτικέ ομάδε για όλη την προσπάθεια που, γίνεται ώστε να που έγινε ώστε να ολοκληρωθούν γρήγορα αυτέ τι διαβουλεύσει. Η Επιτροπή ε, αντιλαμβάνεται ότι για σας τα, οι συμπληρωματικές επεξηγήσεις προκαλούν τουλάχιστον ανάγκη για συζήτηση. Επίσης, αντιλαμβανόμαστε ότι έχετε τους λόγους σας για τους οποίους διατυπώσατε τη μονομερή δήλωση ως ε, έκφραση και ερμηνεία των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυνάμει ε, των συνθήκων δηλαδή και των αρμοδιότητων που έχει ε, από αυτές, αλλά ταυτόχρονα και σε έκφραση πολιτικής βούλης του Κοινοβουλίου. Με το τωρινό πακέτο, αυτά δηλαδή που έχει δεχθεί το Συμβούλιο, αυτά που έχει προτείνει το Κοινοβούλιο, είμαστε στην ενδιάμεση αυτή αναθεώρηση, σε ένα επίπεδο κατώτερο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν σημαντικά βήματα πρόοδου για την υλοποίηση από την περίοδο 2017-2018 και μέχρι το 2020 ε, κατά ευχερέστερο τρόπο των ε, δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, η ενίσχυση της ενσωματωμένης ευελιξίας και μεταξύ των διαφόρων ε, τίτλων του προϋπολογισμού, αλλά και από χρόνο σε χρόνο, γιατί έτσι μπορούμε και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις, νέες δαπάνες και πάντα βέβαια με, με την έμφαση που έχει ορίσει το Κοινοβούλιο με τις προτεραιότητές του. Πέραν της ευελιξίας έχουμε και πρόσθετα μέσα, κονδύλια. Δραστηριο... Έχουμε τη δυνατότητα να δραστηριοποιήσουμε πρόσθετα τα κονδύλια. Ευελιξία λοιπόν, νέα κονδύλια, νέα μέσα σημαντικά για την υλοποίηση των στόχων της καταπολέμησης της ενεργείας κυρίως των νέων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, της εξασφάλισης χρηματοοικονομικής βάσης για την ε, αντιμετώπιση των δαπανών των σχετικών με τη μετανάστευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την υποστήριξη κρατών γειτονικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα οποία προκύπτουν σημαντικέ συνέπειε από τη μετανάστευση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευελιξία και στο κεφάλαιο συμμετοχή, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας μιας πρότασης που θα πάει τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την άμυνα, συγγνώμη. Βρίσκεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ε, στάδιο επεξεργασία μια πρόταση που θα πάει τον Ιούνιο στο Συμβούλιο και θα τη δείτε βεβαίω και εσεί, έτσι ώστε να καταλήξουμε τελικά σε μια εξοικονόμηση πόρων ε, σχετικών με την άμυνα για του 27 αλλά βλέπουμε ότι δεν αρκούν τα κεφάλαια όπως θα προβλέπει ο τωρινό προϋποβολ... Έτσι λοιπόν αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση επιτρέπει να αναπτυχθεί ένα ένας μηχανισμός, μια εργαλειοθήκη για δαπάνες νέες ή ε, προβλεπόμενες μέσα στις οποίες θα έχουμε ένα περιθώριο κινήσεως. Ξέρετε, ότι ήταν πολύ σημαντική και ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ιταλία. Ε, υπάρχει όμως και εξής δέσμευση, ότι παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση στην αγορά εργασίας για τους νέους ε, ανέργους ότι θα παρακολουθούμε την διάθεση των κονδυλίων που προβλέπονται και μέχρι το 2020 ενδεχομένως να χρειαστεί να κινητοποιηθούν νέα κονδύλια για να ενισχυθεί η δυνατότητα των νέων να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας της Ευρώπης. Σήμερα το βράδυ πρόκειται να συναντήσω τον Προεδρεύοντα εκ μέρους της ε, ε, Προεδρίας της Μάλτας και με την ευκαιρία που προσφέρει και η Σύνοδος του Απριλίου πριν από το Πάσχα μέχρι τις 6 Απριλίου θα έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε πιστεύω αυτή την διάμεση ένας θεώρηση από κοινού. Ε, τονίζω για άλλη μια φορά ότι τρέφω κατανόηση για τις επιφυλάξεις και κυρίως σε σχέση με την κοινή δήλωση για την αξιολόγηση της μείωσης του προσωπικού κατά 5%. Το ελεκτικό συνέδριο, θα επισημάνω, έχει προβεί σε μια ανάλυση εδώ, δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με κάτι το καινούριο, ε, το, την Άνοιξη ενημερωνόμαστε πάντα για τις εξελίξεις στον χώρο του προσωπικού όλων των θεσμικών οργάνων. Και επίσης ξέρετε ότι είσαστε εσείς αρχή συναρμόδια για τον προϋπολογισμό. Έχετε μία από τις σημαντικότερες εξουσίες. Επομένως είναι πολύ σημαντικό αυτό να διευκρινιστεί με βάση τις συνθήκες, με βάση την ανεξαρτησία και τις ε, νομοθετικές σας αρμοδιότητες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci, monsieur. πολύ κύριε Επίτροπε. Επομένως, η πρωτοβουλία που μας προτείνουν οι συνεισηγητές είναι ένα είδος ε, αιτιολόγησης κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να έχουμε ένα statement, ε, μια δήλωση, ερμηνευτική των δηλώσεων του Συμβουλίου. Κατά την άποψή σας, ε, δεν θα τεθεί έτσι σε κίνδυνο η συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου, αν κατανοήσα σωστά αυτά που είπατε. Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν για τα ενθαρρυντικά λόγια και για τις διευκρινήσεις. Οπότε πιστεύω ότι θα μπορούμε πλέον να καταθέσουμε τροπολογίες μέχρι την Τετάρτη 22 του μήνα 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών 27 Μαρτίου. Σε μια εβδομάδα δηλαδή. Οπότε 1η Απριλίου στην Ολομέλεια μπορούμε να υποβάλουμε στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, την πρότασή μας για ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου στην Ολομέλεια. Να την υποβάλουμε. Ο κύριος Ντεπρέ θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν συνηθίζεται και τόσο πολύ, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε σχεδόν από όλους ε, με πολύ καλό τρόπο. Εξαιρετική η δουλειά των εισηγητών, ποιοτική δουλειά με επιχειρήματα, πολύ ποιοτική και με μεγάλη δόση φιλοδοξίας. Έπειτα έχουμε μια καλή πρόταση της Κομισιόν. Ε, όταν λάβαμε την πρόταση της Κομισιόν, μπορεί κάποιοι φίλοι, κάπως μαξιμαλιστές και δείτε πώς θα αποκοιτάω, να απογοητεύτηκαν κάπως, αλλά τέλος πάντων υπήρχε μια διάθεση ισορροπημένη και διάθεση να επιτευχθούν πολλά πράγματα με την πρόταση τη Κομισιόν. Μετά είχαμε τη Σλοβάκικη Προεδρία που θεωρούσαμε ότι δεν είναι ιδιαίτερο πεπειραμένη, χρειαζόταν ομοφωνία στο Συμβούλιο. Τι είδαμε όμω, ότι οι Σλοβάκοι σήκωσαν τα μανίκια, ασχολήθηκαν με το θέμα και κατάφεραν σχεδόν την ομοφωνία, κάτι αξιοσημείωτο εκ μέρου τη Σλοβακική Προεδρία που αρχικά δημιουργούσε ανησυχίες σε πολλές αντιπροσωπείε και στη δική μεταξύ άλλων. Και έπειτα είχαμε πολύ καλό ε, suspense εδώ βέβαια αστιεύομαι. Οι σπεσιαλίστες της Κομμέντια Ντελάρτε έπαιξαν ε, το ρόλο τους ε, απόλυτα καλά. Ιταλική επιφύλαξη. Τέλος πάντων, που φτάσαμε ακόμη και αυτοί που ήταν κάπως απογοητευμένοι αρχικά, όλοι ενωμένοι και οι συγητές βέβαια πάνω απ' όλα λένε ότι τώρα μπορούμε να δεχθούμε αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση και αυτά τα έξι δις, τα παίρνουμε τα δεχόμαστε. Για τη δήλωση να κάνω μια δήλωση. Το statement αυτό, για να μην ε, μπερδέψουμε τα πράγματα, είναι πολιτική δήλωση που δεν αλλάζει το δίκαιο, δεν αλλάζει την νομοθεσία. Στη δήλωση του Κοινοβουλίου μιλάμε για τις προνομίες των ε, δύο σκέλων της επί του περιπολογισμού που δεν ε, τροποποιούνται από την πολιτική δήλωση. Κοινή ή μη κοινή. Δεν βλέπω γιατί το Συμβούλιο να πει ότι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα, ενώ το Συμβούλιο έχει δικαίωμα, να δημοσιοποιήσουμε και εμείς σε μία δήλωση, μονομερή, όχι κοινή. Αφού αυτοί το κάνουν, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Και πρόκειται, επαναλαμβάνω, για ερμηνευτική δήλωση στην προκειμένη περίπτωση. Επίση, σε κάποιε περιπτώσει ανησυχούμε. Υπάρχει κρίση νομιμοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε ένα μεγάλο μέρο τη κοινή γνώμη. Υπάρχουν στιγμές που διαρωτώμεθα. Έχουν κατανοήσει όλοι πόσο επίγοντα είναι κάποια ζητήματα. Ότι χρειάζεται κάτι επιγόντως ισχυρότερη ανάπτυξη και μέτρα υπέρ της απασχόλησης των νέων. Μην χάσουμε και τους νέους ε, ύστερα από τα λαϊκά στρώματα. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών τώρα. Δεν μιλώ για υποχώρηση στις πιέσεις μεταναστευτικές, αλλά για αντιμετώπιση αυτών των ε, μεταναστευτικών ε, ροών και αν δεν καταφέρουμε όλα αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίσουμε, θα είναι άσχημα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2019. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Σαρτουή. Σα ευχαριστώ, κύριε Ντεπρέ, που υπενθυμίσετε ότι ε, οι δηλώσει ουσιαστικά είναι κείμενα καλόπιστα από πλευρά ε, όσων υποστηρίζουν ε, την διάμεση αναφέρουσα. Αυτό είναι καλό να το πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι κάθε χρόνο συζητείται ο προπολογισμό ο κύριο Κέλμελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τους δύο συνεισηγητές για πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν θα ήθελα να επισέλθω τόσο σε λεπτομέρειες, ε, διότι μας πιέζει και ο χρόνος. Ίσως όμως θα ήθελα σύντομα σε ό,τι αφορά την ε, μεγαλύτερη ευελιξία. Ε, θεωρούμε πάντοτε είναι θετικό αυτό γιατί πώς λέει το όνομα ε, της λέξης ε, θα είμαστε πιο ευέλικτοι με την διαχείριση των κονδυλίων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγαλύτερη ευελιξία σημαίνει ότι ένα ποσό που έχει οριστεί μία φορά μόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και έχουμε ορίσει τον αρχικό του σκοπό. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ευέλικτοι, σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα που προέρχονται για ένα αρχικό σκοπό, τα αφαιρούμε αυτόν τον αρχικό σκοπό. Αυτό θα πει μεγαλύτερη ευελιξία. Και σε πολλέ περιπτώσει ε, δεν ε, θα λύσει η μεγαλύτερη ευελιξία τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ναι, χρειαζόμαστε συνεχώς περισσότερα χρήματα Εντάξει, μπορούμε να το πούμε. Δεν τα έχουμε όμω ε, στη διαθέσή μα αυτά τα χρήματα και ούτε μπορούν να τα συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη. Δεν να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Μία παρατήρηση τώρα ουσιαστική. Θεωρώ ότι θα έπρεπε ε, στο πλαίσιο της ε, αξιολόγηση ή αναθεώρησης πολιτούς μεσονικού πλαισίου και σε ό,τι αφορά και τι συζητήσει για την κατάσταση του νέου δημοσιονομικού πλαισίου να Είμαστε ξεκάθαροι στη θέση μας ότι δηλαδή εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει ξεκάθαρα να εκθέτουμε τους στόχους μας. Ποιος έχει την ποια αρμοδιότητα και πάνω απ' όλα. Τελικά ποιος είναι έτοιμος να φέρει πιο βάρος. Διότι αν αυτό δεν το κάνουμε μπορούμε να λέμε πολύ ωραία λόγια, ότι θέλουμε να κάνουμε πιο πολλά πράγματα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, για να επιλύσουμε τα προβλήματα της μετανάστευσης. Αλλά επειδή βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το θέμα της μετανάστευσης, βλέπουμε ότι λείπει μια κοινή αντίληψη. Ε, δεν έχουμε μια βάση κοινή ε, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Επίσης, ό,τι αφορά την κοινή αμυντική πολιτική, το επόμενο θέμα, μπορούμε αφαιρετικά να συζητούμε αλλά όταν θα πρέπει συγκεκριμένα μετά να καθαρίσουμε τα πράγματα, ποιος θα είναι αρμόδιος. Ε? αν θέλουμε να έχουμε εξελίξεις ε, ε, στον τομέα της άμυνας, αυτό ουσιαστικά είναι ίσως και αυτονόητο και απλό και δεν χρειάζεται ίσως να το συζητούμε. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βρούμε την απαραίτητη πολιτική βούληση και όχι να συζητάμε για ποσά συγκεκριμένα, για αριθμητικά στοιχεία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε. Ο Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον εισηγητή και τον Επίτροπο Έτιγκερ. Που έδειξε μια κάποια ευαισθησία για τα θέματα που κρίνει άκρο σημαντικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα λόγια του πράγμα το οποίο δεν βλέπουμε να δείχνουν και άλλα θεσμικά όργανα στις Η πολιτική δήλωση λοιπόν του Κοινοβουλίου είναι μια απολύτως φυσιολογική προσέγγιση. Αν δούμε τις δηλώσεις ε, του Συμβουλίου που εγκρίνονται κάθε φορά σε αιτήσει ε, διαπραγματεύσεις και θεωρούνται κάτι το αυτονόητο μέσα από τη διαδικασία της συνθήκης για να έρθουν κάποιες αλλαγές. Αυτό δεν θα έπρεπε λοιπόν να αποτελεί πρόβλημα για μας. Είναι σημαντική η πρόοδος λοιπόν ε, σε μια κατάσταση δύσκολη Όταν οι διαπραγματεύσεις του 2013 ήδη ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία και ήταν ορατή η δυσκολία, η ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε, αντι... είχε έρθει αντιμέτωπη με την Ιρλανδική Προεδρία, με αδυναμία επί έξι μήνες να γίνει διαπραγμάτευση και βρεθήκαμε ενώπιον μιας κατάστασης ότι έγινε συμφωνία ε, για τα διαδικαστικά που οδήγησε, ήταν ταυτόσιμη μια συμφωνία επί της ουσίας και έτσι μπορέσαμε, χάρη και στο συνάδελφο Κάλφιν ε, της ομάδας μου, ε, να κλείσουμε το θέμα μιλώντας όχι για τα χρήματα αλλά για περισσότερη ευελιξία στην, αξιολόγηση, στην αξιοποίηση των κονδυλίων που ξέραμε ότι μέσα στην πρώτη διετία, τριετία δεν θα είχαν ε, τη δυνατότητα να απορροφηθούν. Και έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο για το υπόλοιπο ήμιση της περίοδου. Με κάθε βέβαια επιφύλαξη των όσων θα έφερνε η κρίση στην εξέλιξη της. Η μεγαλύτερη λοιπόν ευελιξία έφερε μια λύση και προσέφερε στο να μπορέσουμε να μετακυλήσουμε κονδύλια σε μια κρίση που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2005 και μάλιστα κατά τρόπο ε, πρωτόγνωρο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι αυτό οφείλει να το αναγνωρίσει και το Συμβούλιο και πρέπει να το ζητήσουμε και για τις προσεχείς δημοσιονομικές προσωπικές ε, προοπτικές να αρχίσουν οι διαπραγματεύσει. Ε, πρόεδρε, όμως ε, πρέπει να πω το εξή ότι ξεκινήσαμε περίπου από μερικούς μήνες ήδη, αλλά δεν έχουμε κάνει αρκετή δουλειά ακόμη. Βλέπουμε την Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον προβληματισμό για τις εναλλακτικέ που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες. Με βάση αυτά που έχουμε να συζητήσουμε, λοιπόν, ε, ω προοπτικέ, πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να τα εκφράσουμε σε μια δημοσιονομική πολιτική. Αν λέμε θέλουμε αυτού του τύπου την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει πάλι να ξέρουμε ξεκάθαρα πώ θα την οργανώσουμε και σε θεσμικό επίπεδο και σε κατανομή ε, πόρων μεταξύ ε, τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου και επίση ποιο θα προσφέρει του σχετικού πόρου. Ιδάλω δεν έχει κανένα νόημα όλη αυτή η συζήτηση. Με τα πιλωτικά λοιπόν ε, προγράμματα όπως αυτό που αναφέρατε τώρα για την έρευνα και την άμυνα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με συνθήκες που δεστιχούν και σε άλλους ε, τομείς πολιτικής. Ε, όταν ανάγουμε ε, μια πολιτική επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς με τα κράτη-μέλη η κατανομή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. Εσείς τι πρόκειται να κάνετε για να οικοδομηθεί εξ αρχής όλη αυτή η νέα δραστηριότητα, η κατανομή των ευθυνών, των καθηκόντων σε σχέση με τα διάφορα υπουργεία που υπάρχουν και που σε ένα βαθμό θα καταστούν στη συνέχεια περιτά, οι αρμοδιαίτες θα καταστούν περιτές καλύτερα. Και αυτό το είδαμε και με την ε, Εξεταστική Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει η Επιτροπή να δρά κατά τρόπο ανεξάρτητο. Έτσι. Έχει λοιπόν την ανεξάρτητη επιτροπή στην εξάρτητη υπηρεσία συγγνώμη, στην Πάρμα. Αλλά υπάρχουν και άλλε εθνικέ υπηρεσίε για τον τομέα των τροφίμων. Ε, το ίδιο μπορούμε να πούμε για κάθε τομέα πολιτική, ότι είμαστε κάπω αμελεί στο να πείσουμε και να εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να αναγνωρίσουν τι ευθύνε του από το η συγκέντρωση εξουσιών που μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υλοποιούνται κατά πιο αποτελεσματικό τρόπο, αλλά που δεν είναι διατεθειμένα να ε, παραχωρήσουν. Το ίδιο και για την αποτελεσματικότητα τη χρήση τη ενέργεια και σε άλλου τομεί. Γι' αυτό λοιπόν για να έχουμε μια σοβαρή χρηματοδότηση πρέπει να εξετάζουμε τι θα έχουμε και τι θέλουμε να έχουμε στο εθνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Πρέπει να δούμε αν ξέρουμε τι περιμένουμε από την Ένωση. Γραμμές πιστώσεων για να εκτελεστούν ε, λειτουργίε που δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη. Καταπληκτικό. Αλλά είναι πραγματικά πολύ ε, καταθλιπτική ως προσπάθεια. Θα γιορτάσουμε την 60η επέτειο από την υπογραφή της συνθήκη της Ρώμης αύριο. Ας πούμε επιτέλους ποια είναι τα προνόμια και αρμοδιότητες του εθνικού επίπεδου. Κυρία Τομά, Αξίζετε. Συγχαρητήρια. Να είστε περήφανοι για όσο έχετε κάνει. Και κύριε Επίτροπε, αυτήν την ε, συνεννόηση πρέπει να έχουμε με το Συμβούλιο όταν θα σκεφτούμε και πώς θα διαρθρώσουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Εξαιρετική δουλειά όντω. Ευχαριστώ όλου όσοι συνεισέφεραν και η Επιτροπή με τις ε, ε, τοποθετήσεις της που εξυπηρέτησε πάρα πολύ και τη δική μας δουλειά και την συνεννόηση μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου για να προχωρήσουμε. Επετέχθη κάτι που δεν ποτέ τώρα δεν είχε γίνει. Δέσμευση για την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για την αναφέρωση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου που ήταν απαραίτητη ως ενδιάμεση και εγκρίνουμε αυτήν την αναθεώρηση. Αυτό δεν θα προδικάσει καθόλου τις αιτήσεις συζητήσεις μας για τον προπολογισμό της Ένωσης. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Θα παραμείνουμε σε αυτά και τώρα θα αλλάξουμε τη σύσταση, θα την κάνουμε μεικτή με τη συμμετοχή της Επιτροπής ΕΚΟΝ με άλλο ένα θέμα πρώτης ε, γραμμής για την παράταση της λειτουργίας του ΕΦΣΥ. Ναι. Bien, comment ça se passe